Right. everybody. I've waited λοιπόν, λοιπόν, αρκετά περίμενα για να έρθουν περισσότεροι σκιώδεις. Για το πρώτο σημείο δεν μπορούμε να περιμένουμε βέβαια ΣΑΗ. Πρώτο σημείο, έγκριση μερισσίας διάταξης. Φαντάζομαι την εγκρίνεται, δεν βλέπω να διαφωνεί κανένας. Ανακοινώσεις της Προέδρου δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Κούτας. Mulțumesc, doamna președinte. Acest raport urmă... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή intervenții ale acesteia, inclusiv obligațiunilor pentru proiecte,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 Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή και γι' αυτό η όλη μου ιδέα θα ήταν ε, να αποφύγουμε να υποβάλουμε τροπολογίες που θα αλλάξουν το αρχικό κείμενο. Καλύτερα να εστιάσουμε στην ε, διατύπωση, αν θέλετε, καλύτερη διατύπωση κάποιων ιδεών που υπάρχουν στην ε, έκθεση αυτή για να γίνουν πιο ολοκληρωμένοι. Και μάλιστα αναφέρομαι σε δύο χαρακτηριστικά. Την εμπλοκή της ΕΤΕΠ στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του να έχουμε πιο καινοτόμε προσεγγίσεις στο χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία εμπλέκουν τους ευρωπαϊκούς ε, τραπεζικούς οργανισμούς όπως την ε, ΕΤΕΠ ή την ΕΤΕ και εδώ αναφέρομαι στην παροχή επιδοτήσεων και δανείων και για να ενισχυθούν τα ε, επενδυτικά κεφάλαια, το venture capitals και επίσης για να υπάρχει ένα μοίρασμα του ανάληψης κινδύνου. Αυτά είναι κάποια χρωμοδοτικά εργαλεία τα οποία κατά θα πρέπει να αναδειχθούν πολύ περισσότερο και να επεκταθούν με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ε, δρομολογημένη χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ είναι η χρήση των ε, δημόσιας χρηματοδότησης για να ενισχυθεί η μοχλευτική ισχύ, για να μπορεί δηλαδή να ενισχυθεί σε συνδυασμό με τον ε, ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο έχει πολύ, πολύ καλό ιστορικό η ΕΤΕΠ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Υπάρχουν τρεις πρωτοβουλίες όπου αυτού του τύπου η λειτουργία, η μοχλευτική των διαρθρωτικών ταμείων μέσω της χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ είναι ε, έντονα παρούσα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου η χρηματοδότηση πολύ μεγάλων έργων υποδομής στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια στα επερχόμενα χρόνια θα αποτελέσουν και τη μείζωνα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δημόσια χρηματοδότηση επομένως δεν θα είναι, δεν μπορεί να είναι η αμυγής και μοναδική λύση. Γι' αυτό χρειάζεται η δημοτική χρηματοδότηση για να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας. Και γι' αυτό υποστηρίζω και εδώ την ε, τροπολογία για τα ομόλογα σχεδίου, τα bonds, ε, project bonds που είναι υπό προετοιμασία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕΠ και που μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν για να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Υποστηρίζω λοιπόν γι' αυτό και τις περισσότερες τροπολογίες που έχουν κατευθεί και θα ήθελα να δω αυτή την μοχλευτική ισχύ να λειτουργεί με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν περιγραφεί και εδώ στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο του θέματος. Πασκάλ. Καλώς απόγευμα. Καταρχάς, κύριε Σιγητά, θέλω να πω ότι η ομάδα των Πρασίνων εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση ως έχει. Υπάρχουν κάποιες ε, περισσότερο διαθετήσει που έχουν γίνει παρά σημαντικέ ε, τροπολογίες που θέλουμε να κάνουμε. Θέλω να τονίσω ουσιαστικά τρεις πτυχές. Η πρώτη αφορά στην αναγκαιότητα κατά όψη μας να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τα κλιματικά κριτήρια και τα θέματα της ενέργειας, την, ενεργητική, ε, την διάσταση ενέργειας. Πρέπει να διευκρινιστεί στην ε, έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος στη χρηματοδότηση της ε, μετάβασης προς την ε, οικολογική προσέγγιση. Ξέρουμε, ακόμα και λόγω συγκυριακών, ε, αν θέλετε λόγων αυτή τη στιγμή, ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου και η Ευρώπη εξαρτάται πάρα πολύ από πηγές εκτός της Υπήρου για την ενεργειακή της τροφοδότηση. Πρέπει λοιπόν η ΕΤΕΠ να είναι ένας καταλήτης, ένας μοχλός για να μπορέσουν να υπάρξουν οικολογικές επενδύσεις οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τους γενικότερους στόχους της μείωσης διοξιδίου του άνθρακα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και και το ζήτημα των επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στις ε, υποδομές ε, των, ε, των εργοστασίων που λειτουργούν με άνθρακα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να μετασχηματίσουμε και να περάσουμε από το ένα μοντέλο στο άλλο μέσα σε λίγους μήνες. Όμως αν γίνει μια διαδικασία phasing out, μια σταδιακής ε, ε, απεμπλοκής ε, από αυτού του τύπου την ενέργεια μέσω χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ, ώστε να μετασχηματιστούν και να αλλάξουν αυτοί οι τρόποι λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών εργοστασίων, θα είμαστε σε καλή πορεία. Ένα τρίτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι να πράξει μια διατύπωση που θα προτάσει τα ομόλογα ε, σχεδίων, τα project bonds και το ρόλο του στο μετασχηματισμό τη Ευρωπαϊκή οικονομίας και επόμενο σημείο σε ό,τι αφορά του φορολογικού παραδείσους. Το αναφέρετε και εσεί στην έκθεσή σα, και αυτό είναι ικανοποιητικό. Θα ήθελα όμω να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι το αίτημα που γίνεται προς την ΕΤΕΠ με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, λέει ότι έχει κάποια πολιτική σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων των χρηματοδοτούμενων, ε, χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων ε, και παρακολούθηση των επενδύσεων σε τόπους ενδεχόμενα φορολογικού παραδούσους, θέλουμε πιο στενή επιτήρηση. Ρωτάμε λοιπόν και θα θέλουμε να ξέρουμε πόσε εταιρείε έχουν αλλάξει έδρα, που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕΠ, Πόσοι εξ αυτών έχουν κριθεί ότι δεν ευθυγραμμίζονται στην πολιτική τη ΕΤΕΠ σε ό,τι αφορά του φορολογικού παραδείσους. Αυτά να έχουμε δηλαδή ένα είδος ανατροφοδότηση ε, των συγκεκριμένων συνεπειών από αυτή την πολιτική που έχει ακολουθηθεί σε σχέση με τους φορολογικούς παραδόσους. Γιατί πέραν των μεγάλων δεσμεύσεων θέλουμε να δούμε και ποιες είναι ο συγκεκριμένος αντίκτυπος των πολιτικών αυτών. Αυτά. Ευχαριστώ. Any... Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κανένας άλλος. Α, ο Ζαν Πολ. Συγγνώμη κυρία, μια συν... σύντομη υπενθύμηση ή θα πρέπει να φανούν, αν θέλετε, όλες ε, οι πολιτικές ομάδες με τις σημαίες τους ή όχι. Αυτή τη στιγμή είναι μια, μια αίθουσα κοινοβουλευτικής επιτροπής και όχι πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν και ζητώ από τους ε, κλητήρες να, βγάλουν τις δύο ε, σημαίες οι οποίες βρίσκονται στο βάθος. I'm sorry, is our group room indeed, but uh, they... συγχωρείτε. Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι ακόμα εκεί. However, Jean Paul, it's Περιπτώσει όμως, Jean Paul, εγώ υποχρεούμε να, τις, να κοιτάω τα πόστερα αυτά, όχι εσύ, άρα είναι ίσω λιγότερα προσβλητικά. Ε, Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν γίνονται πράγματα από την πλάτη μου, εν τούτης θα αισθάνομαι και τα καταλαβαίνω. Eyes in the back of your head. That's uh, very... Κατάλαβα. Έχεις μάτια και πίσω στην πλάτη. Πολύ καλό αυτό για να συντονιστεί. Λοιπόν, εάν θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Ούτω. για να αυτό στην παρατήρηση του Ζων Πολ. Θα μπορούσε ίσως αναλεκτική να προτείνω όταν ξανασυνεδριάζουμε στην αίθουσα των φιλελευθέρων να έχουμε τόσα πλακά όσα μέλη έχουμε στην ομάδα μας από τους φιλελεύθερους να το λάβουν υπόψη μας. Γιατί βέβαια οι φιλελεύθεροι ο καθένα έχει τη δική του μεμονωμένη θέση. Ε, εντάξει, τούτο λεφθέντος ε, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σοβαρότητα τη έκθεσης του συναδέλφου και φίλου Κούτας. Ε, το τη συζήτηση δεν θα πρέπει να μας κάνει να παραβλέπουμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δούμε πώς θα ε, συμβάλλουν τα μέσα αυτά στην ε, πολιτική καταπληκτική κρίση. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο Κούτας και να καλέσω όλους τους συναδέλφους να συνεργαστούν επικοδομητικά. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ και έχετε το λόγο. Okay. To do with the um, project bond όσον αφορά αυτά τα project bonds, τα ομόλογα σχεδίων που αναφέρθηκαν από διάφορα μέλη. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε πάλι μια σύγκρουση δύο επιτροπών, γιατί η προσωρική, προσωρινή έκθεση κρίσης συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και εξτάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Και πραγματικά θα ήθελα να πω εκεί να μπορέσω να συζητήσω, να ακούσω τις λεπτομέρειες συμμετέχει η Κομισιόν εκεί. Είναι πραγματικά ε, κακό σημαντικό ότι κάτι που έχει επιπτώσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και που μα αφορά όλους εμάς για τη μελλοντική χρηματοδότηση για τα διάφορα σχέδια είναι αντικείμενο αυτή τη σύγκρουση των συμφερόντων. Όλοι θα διαβαράμε να ακούσουμε τι λέγεται και δεν ξέρω πώ μπορεί να λύσει αυτό το θέμα. Πολλοί από εμά είμαστε και στι δύο επιτροπέ ε, και προτιμήσαμε να έρθουμε εδώ επειδή είμαστε συντονιστέ. Αλλά ήταν καλό να μπορούσαμε να είμαστε ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Θα ήθελα επίση, η Επιτροπή να έχει μια σοβαρή συζήτηση εκτός από την ετήσια έκθεση της, ε, του θέματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημαντική απόκριση από το παρελθόν όσον αφορά τη χρηματοδότηση και πολλά από αυτά θα ασχοληθούν με συγκεκριμένα μέσα, αρχήματα και ε, το τι θα χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις κλπ αυτά τα προτείνουν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε αναλυτική συζήτηση του θέματος. Μέχρι σήμερα εγώ νόμιζα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ήταν εκείνη που θα εκδώσει αυτά τα ομόλογα. Αλλά από το έγγραφο που μόλις διάβασα υπάρχει φαίνεται μια νέα μονάδα που αναφέρεται σαν μια πρωτοβουλία με κεφαλαίο π, δηλαδή υπάρχει κάτι που κρύβεται, κάποιος οργανισμός. Δεν ξέρουμε όμως ποιες είναι λεπτομέρειες. Μήπως θα πει η πρόεδρος να μας βρει όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να μας τις μεταβιβάσει εδώ στην Επιτροπή μας. Πρόεδρος, φυσικά, είναι κάτι το οποίο ανέφερα ήδη σε άλλο πλαίσιο. Έχουμε εδώ Αλεξάνδρ Καραμένου. Δεν ξέρω, θα μπορέσει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες συμπληρωματικές. Thank you very much, Mrs. Chair. Uh σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο των ε, ομολόγων σχεδίου, όπως ξέρετε σήμερα δρομολογήσαμε την ε, δημόσια διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος μας έχει προσκληθεί να μιλήσει στην ε, Επιτροπή σου αργότερα πάνω σε κοινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σίγουρα θα ήθελε ευχαρίστω να έρθει εδώ αν το επιθυμείτε τις επόμενες ημέρες για να κάνει την αντίστοιχη παρουσίαση και να συζητήσει μεγαλύτερη λεπτομέρεια το θέμα αυτό. Επιτρέψτε κάποιε ε, πιο συγκεκριμένε παρατηρήσει. Τα ομόλογα αυτά δεν εκδίδονται ούτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτε από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Εκδίδονται από ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίε είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή, ε, εκτέλεση των έργων αυτών υποδομή. Εξετάζουμε την πιθανότητα χρησιμοποίηση του κοινοτικού προϋπολογισμού και των μηχανισμού της ΕΤΕΠ για να υπάρξει εγγύηση των ομολόγων αυτών για να μπορούν να υπάρξει έλξη ιδιωτικών ε, κεφαλαίων. Δεν είναι δηλαδή μια έκθεση ομολόγων από Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων ή από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαρίστως να σας ε, παράσχουμε και συγκεκριμένο γραπτός, ε, αν θέλετε, μια περιγραφή των εργαλείων αυτών, να σα δείξουμε τι ιδέε που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμή στην Επιτροπή, ε, βέβαια κατανοώντας σε απολυπεράς ότι πρόκειται για ενεξελίξη εργασία. Τώρα, σε κάποια άλλα σημεία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Κούτα, για την εξαιρετική του εργασία και όλους τους άλλους που έχουν συνεισφέρει στις τροπολογίες. Είναι ευπρόσδεκτες από πλευράς μας σε σχέση με τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πληροφοριακά σας λέω ότι μόλις δημοσιεύσαμε τα ετήσια στοιχεία μας ό,τι αφορά το 2010, και η συνολική χρηματοδότησή μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τον στόχο ο οποίος είχε καταρτιστεί ε, σύμφωνα με το ε, σχέδιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανασυγκρότησης των 30 δις του 2008. Έχουμε, αναπτύξει, έχουμε θεσμοθετήσει, έχουμε συντάξει ένα νέο νόμο για τις ε, ε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 2009 που αφορά στις χώρες που είναι προσένταξη και που ήδη συμπεριλαμβάνει στοιχεία μεγαλύτερης διαφάνειας και μεγαλύτερης δέσμευσης από τους ε, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβούντες ώστε να περάσει μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει και δέσμευση από τους διαμεσολαβητές να μπορέσουν να συγκεράσουν την ε, κοινοτική χρηματοδότηση με, από την ΕΤΕΠ με αντίστοιχη ιδιωτική χρηματοδότηση. Έχουν καταβληθεί λοιπόν ήδη σχετικέ προσπάθειε και με την ε, προσφορά και τη συνδρομή του Κοινοβουλίου μπορούμε να πετύχουμε περισσότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις χώρους εκτός δικαιοδοσίας, δηλαδή τις εταιρείες, αν θέλετε, τους χώρους offshore. Έχουμε ήδη αναπτύξει νέες πολιτικές το 2001, που θεωρήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι, αν θέλετε, πραγματικά στον ε, ε, να είναι πολύ προθυμένες σε ό,τι αφορά ε, τις διαδικασίες αυτές και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία διασύνδεση είτε κάποιου χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή ή αντισυμ, οικονομικού αντισυμβαλόμενου να έχει σχέση με εταιρείε offshore. Υπάρχουν κατάλογοι οι οποίοι έχουν συνταχθεί από άλλους διεθνείς οργανισμούς τέτοιων offshore εταιριών. Δεν υπάρχει επίσημος βέβαια κατάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να βασιστούμε στους καταλόγους άλλων ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών. Δεν έχουμε δηλαδή δικό μας κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Βασιζόμαστε στον κατάλογο που έχει εκδώσει ο ΩΣΑ ε, κλπ. Τώρα, κάτι μικρό που αναφέρθηκε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο κλπ. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την νομοκλευτική ισχύ που αναφέρθηκε, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα ενίσχυση αυτή τη νομοκλευτική ισχύω, ε, ώστε να γίνει καλή, χρήση των κοινοτικού προπολογισμού και των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων και κρατώντα την, ε, την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα τη ΕΤΕΠ, δηλαδή 3α, που είναι ζωτική σημασία για να μπορέσει να προσελκύει ιδιωτικά κεφάλαια και να ε, διαβιβάζει, αν θέλετε, και να μεταβιβάζει το οικονομικό αυτό όφελο προ του ε, πελάτε μα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και άλλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα σημείο το οποίο μόλις ε, σκέφτηκα, είπες ότι για την η ΕΤΕΠ δεν θα εκδίδει, αλλά θα είναι εγγυητή των ομολόγων αυτών. Άρα το ερώτημα είναι πού θα εμφανίζεται αυτή η εγγύηση στον ισολογισμό της ΕΤΕΠ θα συγκρίνεται με τον τρόπο που ε, ελέγχονται τα κράτη-μέλη από τη Eurostat ότι θα πρέπει να εγγράφουν στους ολογισμούς τους όλες τις σχετικές εγγύησεις που έχουν ε, εγγράψει μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου. Ίσως θα, πρέπει να, θα θέλετε να επανέλθετε σε αυτό. Αλλά συνδέεται με την παρατήρηση που κάνατε σε ό,τι αφορά τους ολογισμούς. Και δεν είμαστε και οι δήμονες επί του θέματος και δεν θα θέλαμε να το δούμε ακριβώς έτσι. Ναι, με την άδειά σας θα απαντήσω. Θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία αυτά στον ισολογισμό. Όλες αυτές οι εγγύησεις θα υπάρχουν στον ισολογισμό της ΕΤΕ και του κοινοτικού προπολισμού έμεσα. Όπως υπάρχει ήδη στον ισολογισμό για τις προβλέψεις των επενδύσεων αυτών. Λοιπόν, και στον προεπλογισμό στο δικό μας και τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ποιο θα ήθελε να επανέλθει, ο εισηγητή. Καταρχήν ευχαριστώ τους συναδέλφου για την υποστήριξή τους και τις ιδέες που παρουσίασαν εδώ. Όσον αφορά την ιδέα να έχουμε μία συζήτηση για το ομόλογο σχεδίων είναι πάρα πολύ καλό. Θα ήταν καλό να καλέσουμε ίσως τον κύριο Μάισταρ να γίνει συζήτηση εδώ, στην Επιτροπή μας και να διευκρινιστούν διάφορα στοιχεία όσον αφορά τις εγγυήσεις, τα σχέδια που θα χρηματοδοτούν κλπ. Και μέχρι αύριο στις 10 θα περιμένω για να συζητήσουμε στους ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. όπω είπατε, οι ψηφοφορίε θα γίνουν τη 15η Μαρτίου και θα περάσει από την Ολομέλεια στον ε, Απρίλιο. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στους ε, χρηματοπιστωτικούς ομίλους και θα δώσω το λόγο στον συντάκτη κύριο Στολογιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω όλους όλα τα μέλη της Επιτροπής που παρουσίασαν τροπολογίες της, ε, στην έκθεση. Πρόκειται για καλές τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, σύμβουλό μου κύριο Βάινες για την συμβολή του κατά την ανάλυση των λόγων τροπολογιών. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πολλές από τις προτινόμενες τροπολογίες με βρίσκουν σύμφωνο. Ορισμένες εξ αυτών εστιάζουν σε ένα καλύτερο ορισμό κάποιων σημείων του εγγράφου της Κομισιόν. Δεν θα επιμείνω επί τροπολογιών φυσικά τις οποίες ε, και στηρίζω, αλλά θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα αναφορικά με πολλές τροπολογίες που χρειάζεται να συζητηθούν αφενός εδώ, αλλά και να συζητηθούν αργότερα με τους εκπροσώπους ε, τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και του Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα αφορά τον προσδιορισμό του κατά πόσον οι δραστηριότητε ενός ομίλου έχουν σχέση με τον ε, χρηματοπιστωτικό κλάδο και εδώ έχουμε τροπο, τροπολογίε τροπολογίες, 92 παραδείγματο ε, της Λάμπερτ, του κυρίου Λάμπερτ συγγνώμη, και 93 της κυρίας Μπόλφ. Ο κ. Λάμπερτ ε, προτείνει να έχουμε ένα όριο κατόφλι 10 ατόμων. Εάν ε, η οικονομική δραστηριότητα ξεπερνάει το 10% του των ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων οντοτήτων από τον, του συνολικού προπολογισμού τότε τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί ως ε, χρηματοπιστωτικός κλάδος που ανήκει στον Όμιλο. Ε, η κυρία Μπόλ προτείνει ένα ποσοστό 40% και επιπλέον θα πρέπει να μπορούν οι εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές να αποφασίζουν πως το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τραπεζικό κλάδο, στον ασφαλιστικό κλάδο και στους επενδύσεις είναι ουσιώδης. Νομίζω πως η πρόταση της κυρίας Μπόλσου ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάγκη προσδιορισμού αυτής της δραστηριότητας στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους και φυσικά θα την προτείνουμε την πρόταση αυτή. Την υποστηρίξουμε, λοιπόν, την τροπολογία 93. Ένα δεύτερο ζήτημα άπτεται μισό λεπτό να δω για τις μη ρυθμιζόμενες ε, χρηματοπιστωτικές οντότητες ε, τότε ο ισο, ισολογισμός θα πρέπει να υπόκειται σε μια αυξημένη υποπτία. Αυτό αφορά στην τροπολογία 110 του κυρίου Λάμπερτ και Συμφωνώ με τις ανησυχίες του κυρίου Λάμπερτ αναφορικά με τις μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες ε, περιλαμβανομένων των μηχανισμών εκτός ισολογισμού. Λοιπόν, αυτό που τίθεται εδώ είναι να επανέλθουμε στο πεδίο εφαρμογής αυτής της ε, οδηγίας και υπενθυμίζω πως υπάρχουν δύο φάσεις, δύο στάδια. Προκειμένου να τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος ε, των ε, χρηματοπιστωτικών οντοτήτων, ε, ομίλων. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ισχύουσες οδηγίες και τις επιπτώσεις τους επί άλλων οδηγιών αλλά και τις ε, επιπτώσεις τους σε μια νέα οδηγία που αφορά τις ευρωπαϊκές υποπτικές αρχές. Θεωρώ ότι το να εδώ το ζήτημα των μη θυμιζόμενων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων περιλαμβανομένων των μηχανισμών εκτός ολογισμού σε αυτό το ε, σχέδιο οδηγίας καθιστά τα πράγματα περίπλοκα, διότι δεν γνωρίζουμε την αντίκτυπο αυτών των προτάσεων και κρίνουμε πως είναι καλύτερο να κριθεί η εν λόγω πρόταση σε μια δεύτερη φάση όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια πλήρη ανάλυση των αλλαγών που χρειάζεται να γίνουν κατά την, ε, τον έλεγχο των ε, χρηματοπιστωτικών ομίλων και όταν θα φτάσουμε στον ε, μελέτη αντικτύπου. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που αφορά τα, τους διαχειριστές των εναλλακτικών ταμείων εδώ νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Αυτά τα εναλλακτικά ταμεία λοιπόν, που μπορούν, επενδυτικά ταμεία, που μπορούν να ενταχθούν στον τομέα των ε, υπηρεσιών ή σε ένα άλλο οικονομικό κλάδο και υπάρχει πρόταση μπάλς ότι δηλαδή θα πρέπει τα διαχειριστές αυτών των ταμείων να ενταχθούν στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή κατά πόσον αυτά τα διαχειριστές ελαστικών ταμείων εργάζονται για έναν και μόνο κλάδο, τότε θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτόν τον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Αλλά έχουμε και κάποιες καλές προτάσεις ε, σχετικά με ένα ζήτημα που αφορά τα stress test, ε, της δοκιμές αντοχής. Ο εισηγητής και ο κύριος Μπαουλς και ο κύριος Σκίνερ στις τροπολογίες τους αναφέρονται σε αυτά τα stress test και συμφωνώ με τις προτάσεις αυτές Έχουμε ήδη ένα συμβαστικό κείμενο και πιστεύω πως όταν θα συζητήσουμε αυτό το συμβαστικό κείμενο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε προκειμένου να, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλων αυτών των τροπολογιών. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα, κυρία Πρόεδρε, που ήθελα να θίξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, σημείωνα. Right, you're there. <laughs> Sorry. <laughs> I'm losing track of you, Edward. Α, σας έχασα. Πού είσαστε? Α, εδώ ήσασταν. Ναι, εγώ θα σας παρουσιάσω ότι έχω να πω εξ ονόματος του Πίτερ Σκίνερ, που δεν μπορεί να είναι παρόν. Ο Πίτερ χαίρεται για το ευρύ φάσμα των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμε. Συμπληρώνουν τι βασικέ προτάσει του εισηγητή. Λείπει βέβαια ότι ορισμένε αυτέ ίσως ε, παρεξηγούν κάποια στοιχεία. Δεν έχουν ακολουθήσει σωστή γραμμή. Τρία σημεία ακολουθούν οι τροπολογίε. Το ένα είναι να διευκρινίσουν το ρόλο τη κοινή επιτροπή. Εξασφαλίζουν οι ευθύνε τη να είναι ευθυγραμμισμένε με του πόρου και με το νομικό καθεστώ τη και να εξασφαλίζει βασικέ γραμμέ ευθύνη λόγω του διαδοματικού χαρακτήρα των, ε, των ομίλων. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ότι μέσα στους ομίλους αυτούς υπάρχουν νομικές μονάδες και πώς σχετίζονται με την νομική δομή στην οποία λειτουργεί ο ομιλευτή. Και υπάρχουν εδώ τροπολογίες για την ρευτότητα για να υπάρχει και ένα ίσο πεδίο παιδής. Τρίτον, τονίζει τον κανόνα που απογορεύει τις τράπεζες ομίλους να εκθέτουν πάνω από 3% του επενδυμένου ε, κεφαλαίου σε απώλειες από τις επενδύσεις αυτές. Και δεύτερον, αφορούν ένα κενό του κοινωτικού κανονισμού για τις χρηματοπιστωτές υπηρεσίες όσον αφορά αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις. Προσβλέπει να διαπραγματευτεί με τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές για να υπάρχει μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου πριν από τον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης για την ομάδα των φιλελευθέρων. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου λοιπόν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Και όσον αφορά την δική μου 93, ο στόχος ήταν μέσα στα πλαίσια μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να υπάρχει ένα σημαντικό υψηλό κατόφλι. Προσπάθησα λοιπόν να το αντιμετωπίσω αυτό, γιατί το 10% του κατοφλίου είναι σημαντικό. Προσπάθησα λοιπόν να εντάξω κάποια στοιχεία για να είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδοθούν και που θα ακολουθηθούν. Γιατί αλλιώς δίνουμε ίσως μια εσφαλμένη ε, εικόνα των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζών και Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Και έτσι έχουμε τώρα μια άλλη βάση για να ληφθούν αποφάσεις. Στην τροπολογία μου είναι 96, όπου λέω ότι θα πρέπει οι εταιρείε διαχείριση περιουσιακών στοιχείων να είναι πιο πλησίων τη ε, οδηγία και των κατευθυντήριων γραμμών. Φοβούμαι ότι αυτή η τροπολογία κάπως πλησιάζει την ε, τροπολογία 95 του Μπόικα που αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Αν εξετάσει κανένας όλο το στοιχείο αυτό, με την έννοια του πελάτη, με την ευρύτατη έννοια του, του όρου, μπορούμε εγώ να φτάσουμε αυτό. Και για τις κατευθύνες γραμμές, η τελευταία μου τροπολογία είναι 111, όπου αφορά στις εταιρείε που ε, έχουν στα, χέρια τους αυτές τις, ε, τις, ε, αυτές τις μετοχές Νο, θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό και γι' αυτό θα έπρεπε να το διευκρινίσουμε τώρα και όχι να περιμένουμε αργότερα. Θα πρέπει γενικά να δούμε τι γίνεται με τις εταιρείες αυτές των χρηματοπιστωτικών μετοχών. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που μπορούσα να υποστηρίξω, αλλά υπάρχουν και άλλες που δεν μπορώ να υποστηρίξω. Αυτή τη στιγμή νομίζω θα αρκούσε να σας πω ποιο ήταν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχω στηρίξει οι δικές μου τροπολογίες. Φίλιπ Λάμπερτ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς απαντώ στον εισηγητή πάνω στο θέμα των μη ρυθμιζόμενων ε, χρηματοοικονομικών οργανισμών. Από ό,τι μα λέτε είναι ότι δεν είναι του παρόντο, πρέπει να το αφήσουμε να το εξετάσουμε αργότερα. Νομίζω καλό θα ήταν να το αναφέρουμε, ακόμα και αν θεωρείται αυταπόδεκτο, ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλουμε σε μια αιτιολογική σκέψη ή άρθρο, αλλά δεν βλέπω γιατί δεν πρέπει να συμπεριληφθεί. σω πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ελπίζω ότι κανείς ημών δεν υπερασπίζεται ότι θέλουμε να κρατήσουμε αυτούς τους χρηματοοικονομικούς ομίλους εκτός διευθέτηση και κανονισμού. Αυτό το οποίο με εκπλήσει και θέλω να κατανοήσω λίγο την αντίδρασή σας είναι ότι δεν ήμασταν τόσο φιλόδοξοι, τόσο ρισπαστικοί αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τον, ε, αν θέλετε, κατακαιρματισμό των δραστηριοτήτων αυτών των μεγάλων χρηματοοικονομικών, ε, χρηματοοικονομικών ε, ε, ομίλων. Να βάλουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ενδιάμεσα στεγανά ώστε να μην βουλιάξει όλο το σκάφος αν υπάρχει πρόβλημα, να υπάρχουν ενδιάμεση φραγμοί. Στο ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε μη σωστές ή και περιτές μεταφορές κονδυλίων από μια εταιρεία στην άλλη σε τέτοιου είδους μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες προτάσεις πάνω στα συστημα... στους συστημικά πολύ σημαντικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα σχετικά και ξέρουμε ότι κάποιοι από τους οργανισμούς που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μεγάλοι όμιλοι μετά την κρίση και απλώς και το μέγεθός τους και μόνο τους καθιστά ουσιαστικά αδύνατο να παρακολουθηθούν ε, από πλευράς υποπτικής αρχής, ε, είτε εθνικής είτε ευρύτερη υποπτικής αρχής. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταδείξουμε να υποδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, ίσως αν θέλετε όχι τα ριζοσπαστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αποθαρρύνοντας το πολύ μεγάλο μέγεθος τέτοιου είδους ε, χρηματοοικονομικών ομίλων ε, χρηματοπιστωτικών ομήλων, ίσως ε, επιβάλλοντας πολύ μεγάλη κεφαλαιακή απέτηση. Βάλαμε το κατόφλι στα 100 δις. Ίσως θα πρέπει, θα θέλατε να το κάνετε λιγότερο αν θέλετε έτσι ασπρόμαυρο να υπάρχει μια διαβάθμιση, αλλά να υπάρχει κάποια διατύπωση όπου θα μπορούμε να πούμε ότι όντως θέλουμε να αποθαρρύνουμε τόσο μεγάλη μεγέθη. Γιατί από κάποια άποψη το μέγεθος ουσιαστικά και οικονομικά δεν είναι ε, βέλτιστο και προκαλεί και στρέβλωση της αγοράς, γιατί πάνω από κάποιο όριο, κάποιοι οργανισμοί, σκέφτομαι κάποιες πολύ μεγάλες τράπεζες, όπως και ευρωπαϊκές, όχι μόνο βαρύνουν με το μέγεθος αυτού και καθοδηγούν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική αγορά, αλλά και απομακρύνουν και αφαιρούν ε, κύκλο εργασιών από άλλες τράπεζες. Αν δείτε πώς, ε, εμπορεύονται τις κινητές αξίες οι τράπεζες ή τα χρηματιστήρια, θα σκεφτείτε αν θέλετε ότι είναι ουσιαστικά η ιστορία της Microsoft, η οποία καταβρόχθησε ουσιαστικά όλες τις εταιρείες λογισμικού, οπότε η Microsoft έγινε ε, πράγματι ουσιαστικά μονοπόλιο, μια οντότητα που προσφέρει τα πάντα. Αυτό δεν είναι καλό για την αγορά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ. Και αν δεν το κάνουμε, αν θέλετε, εδώ με συγκεκριμένε κατευθύνσει, τουλάχιστον σε θεολογικέ σκέψει, θα πρέπει να υποδεικνύουμε στην Επιτροπή προ τα πού θέλουμε να κινηθούμε. Ευχαριστούμε. Κέιτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο εισηγητή ε, και ο Σκιώδη έχουν καλύψει πάρα πολλέ από τι παρατηρήσει που θέλω να κάνω. Ε, Συνεχίζοντα όμω τα σχόλια που μόνο ακούστηκαν, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και να θυμόμαστε ότι πρόκειται για, μεγάλους για χρηματοπιστωτικού ομίλου. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα πάρα πολύ μεγάλοι, αλλά έχουν ένα μείγμα οικονομικών δραστηριοτήτων που του τάσει κάτω από την οδηγία αυτή. Δεν θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένη δουλειά, που κατακλείδη αν θέλετε συνιστά ίσον αλλαγή παρά ε, θεμελιώδη αλλαγή. Δεν θα ήθελα να αποθαρρύνουμε, αν θέλετε, να θέσουμε ε, σε δυσχερή θέση τις εταιρείε αυτές, του ομίλου αυτούς που εμπίπτουν σε αυτή την περιγραφή έναντι άλλων μεγάλων, αν θέλετε, τραπεζών ή ασφαλιστικών οργανισμών που όντως εξορισμού εμπίπτουν εδώ πέρα. Ε, σε εμά, μιλώντα από, το από το Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο ένα από του ε, οργανισμού μα ε, μπορεί να ενταχθεί, αν θέλετε, να υπαχθεί σε αυτή την περιγραφή που δίνεται εδώ πέρα σε ό,τι αφορά την, ε, το χρηματοοικονομικό όμιλο. Ε, πέραν, αν θέλετε, τραπεζών. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλε τι τράπεζε και όλε τι ασφαλιστικέ εταιρείε σε, σε όλα τα κράτη. Δεν νομίζω ότι ο κίνδυνο είναι διαφορετικό. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικά εργαλεία εκτό ισολογισμού ή όταν εμπλέκεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει διαφορά δηλαδή σε ό,τι αφορά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο για μεμονωμένε τράπεζε, ασφαλιστικέ εταιρείε ή συγκεκριμένη περίπτωση όπω εξετάζουμε εδώ πέρα του ομίλου δεν έχουμε βάλει στις μεμονωμένες χρηματοπιστωτικές ε, οντότητες, τράπεζες ή ασφάλειες τέτοιου είδους περιορισμούς. Άρα δεν νομίζω ότι είναι σωστό να τους βάλουμε εδώ πέρα στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Πρέπει να είναι ισότιμο το παιχνίδι. Μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανησυχία. Εάν βάζουμε τον κανόνα Volcker για τους ομίλους αυτούς, γιατί τους βάζουμε και στις μεμονωμένες τράπεζες γιατί να παίρνουμε μόνο ένα υποσύνολο και όχι ολόκληρο το πεδίο. Οπότε έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όντω εφαρμόζουμε τι ίδιε αρχέ και του ίδιου κανόνε παντού. Προβληματίζομαι επίση, παρακολουθώντα και κάποιε από τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί και που τι ε, διέτρεξα, ότι ερχόμαστε λίγο σε κάπω ε, ποσοστά που είναι αυθαίρετα κατόφλια. Και αυτό λίγο, αν θέλετε, ε, με προβληματίζει, ότι ίσως δεν τα ε, αποτιμούμε ανεξάρτητα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι σχετικό το κάθε κατόφλι. Και δεν νομίζω ότι εμεί ε, ω βουλευτέ ε, είμαστε οι δήμονε και μπορούμε κατά πόσον το 10, 15, 30 ή οποιοδήποτε τη εκατό, οποιοδήποτε νούμερο είναι το κατάλληλο κατόφλι. Θα πρέπει, αν θέλετε, επιστημονικά να αποτιμηθεί. Και η κατόφλι, αυτό θα πρέπει να οριστεί από την συνολική εποπτική αρχή, όχι από εμά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί ότι γενικά θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει ξεχωριστή μεταχείριση για τις οντότητε αυτέ επειδή είναι χρηματοψηφιακοί όμιλοι, θα πρέπει να εξετάσουμε τον κίνδυνο τον οποίο παρουσιάζουν. Εάν ο κίνδυνο ε, είναι μεγάλο σίγουρα, αν θέλετε, δεν θα αφορά μόνο στου χρηματοψηφιακού ομίλου, αλλά σε ολόκληρο το χρηματοοικονομικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι οντότητε αυτέ που αποφασίζουν να έχουν ετερογενεί δραστηριότητε, να έχουν και τραπεζικέ δραστηριότητε και ασφαλιστικέ. δεν θα πρέπει να τι αποθαρρύνουμε ή να τι θέτουμε αν θέλετε σε μειονεκτική θέση σε σχέση με του άλλου ομιλού που αποφασίζουν να έχουν αμυγό είτε τραπεζική είτε ασφαλιστική λειτουργία. Ευχαριστούμε. Ο κ. Σκρούτν δεν είναι εδώ. Ο κ. Λάμπερτ και πάλι τον λόγο εντάχει. Υποθέτοντα ότι θα δώσετε μια απάντηση που θα βοηθήσει. Uh, θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει μόνο ένας οργανισμός ΙΤΑΒ που εμπίπτει σε αυτή την νομοθεσία για να πω ότι ήδη η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει κάποιες, κάποιους ομίλους όπως Μπάρκλε, τον ομίλο Μπάρκλες και, και τους θεωρεί ως ομίλους. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κάποιον ορισμό ιδιαίτερα ευρύ. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Όχι επειδή ε, ενδεχόμενο υπάρχει και ένας ε, συστηματικός κίνδυνος, ε, συστημικός κίνδυνος, συγγνώμη, και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνο τον νόμο για τους ομίλους, μπορούμε να τον εφαρμόσουμε και πρέπει να τον εφαρμόσουμε για όλες τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι τα σχόλιά σας σχετίζονται με τα δικά μου, διότι αν δείτε τις μου, πραγματικά συμπίπτουν τα λεγόμενά σας. Να πω ότι η τροπολογία μου 111 είναι μια πολύ σημαντική τροπολογία και ε, επιθυμεί να αποφύγει την διπλή εποπτεία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχει στήσει κανείς το λόγο, γι' αυτό δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρθηκαν ε, και που αφορούν τον κύριο Σκίνερ το αφορά τον ρόλο της ε, Κοινής Επιτροπής θα πρέπει να το εξετάσουμε μιλάμε για τον νομικό ρόλο διότι αυτή η αρχή δεν έχει την εξουσία να λάβει αποφάσεις και θα δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μέσα στο σχέδιο της οδηγίας αυτή η πρόταση. Δεν έχω καμία ένσταση σχετικά με την διαφάνεια των εκθέσεων. Τώρα αναφορικά με τον κανόνα Βόλκερ θα πρέπει να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε, διότι για μια ακόμα φορά δεν είμαι τόσο υπέρ της ε, υποστήριξης τροπολογιών για τις οποίες, για τις οποίες δεν έχουμε ακόμα μία ε, μελέτη αντικτύπου. Και αυτό δεν αφορά μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά επανερχόμενο στα σχόλια του κυρίου Λάμπερτ και τον ευχαριστώ για τις τροπολογίες. Τροπολογία 114 προτείνει το κατόφλι εάν το συνολικό ισοζύγιο ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και ο λόγο των ομιλούς όμιλου των δραστηριοτήτων δεν μειώσει εντό έτου τον ισολογισμό του εντό των ΟΤΑ του ορίου, υπόκειται σε κεφαλαϊκέ απαιτήσει τριπλάσιε του ποσού που ορίζεται η σχετική νομοθεσία που εμφαίνεται στο άρθρο 1. Κοιτάξτε, ούτε εδώ υπάρχει μελέτη αντικτύπου. Νομίζω πως αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά στην Κομισιόν, δηλαδή στην επόμενη φάση να προβεί σε αξιολόγηση και να μας υποβάλει την αξιολόγηση αντικτύπου προκειμένου να αποκρισταλώσουμε άποψη στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ 100% με όσα υπόθηκαν ότι δηλαδή δεν είμαστε αρμόδιοι, αρμόδιοι να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο κατόφλι εδώ στην Επιτροπή μας, δίχως να έχουμε προηγούμενη να συζητήσει την μελέτη αντικτύπου. Θα συζητήσω με τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες έτσι ώστε να καταλήξουμε κατά το δυνατόν σε συμφωνία και συμβασμό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα προσβλέπουμε μάλλον σε αυτό το αποτέλεσμα. 21-22 Μαρτίου θα ψηφιστεί η έκθεση και στην Ολομέλεια θα περάσει τον Μάιο. Και τώρα που να περάσουμε στο σημείο 5 της Μεσαίας Διατάξεως που αφορά τις ε, τεχνικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Η κυρία Εσάια έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ε, πρότεινε την, ε, έκανε την πρότασή της στις 16 Δεκεμβρίου 2010 πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και συμπεριλαμβάνει ένα και αναφέρει μάλλον τις ε, τεχνικές ε, αυτές απαιτήσει ε, τώρα. Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς θα έχει θετικότατες επιπτώσεις, αύξηση του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και θα μειώσει το κόστος για τους πολίτες, για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Μελέτη εντεκτή που αναφέρει πως τα πιθανά ωφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να ανέρθουν σε 300 δις ευρώ μέσα σε μια εξαετή περίοδο. Τρεις ε, προτάσεις έχουν γίνει και θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση αποτελεί μια πολύ σημαντική πολιτική πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, μεταφορές για τις, πιστές, για τις μεταφορές ε, πιστώσεις και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και τροποποίηση του κανονισμού που γίνεται σε συντονισμό με τα εποπτικές αρχές ε, των ε, τραπεζικού κλάδου. Στις 28 Ιανουαρίου 2008 ξεκίνησε αυτό το σύστημα των μεταφόρων πίστοσης Πάντως η μετάπτωση στο νέο σύστημα καθυστέρησε ιδιαίτερα τον Οκτώβριο 2010, δύο χρόνια μετά από την ε, σύσταση του συστήματος, οι μεταφορές πίστοσης ε, ανέρχονταν σε 9,3%. Και θα ήθελα να πω ότι η τρέχουσα κατάσταση δημιουργεί αβεβαιότητες σε όλους τους ενδιαφερομένους και ιδιαίτερα δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι προέβησαν άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές. Αυτή είναι και άποψη του Κοινοβουλίου, διότι θα ενθυμίσετε πως το Κοινοβούλιο δις ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προωθήσει τον σχετικό κανονισμό. Λοιπόν, τόσο το 2009 αλλά και το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε και παραθέτω πως χρειάζεται μια σαφής ε, πρόταση όχι αργότερα μετά από 31 31η Δεκεμβρίου του 2010 προκειμένου να γίνει η μετάπτωση ολική. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν αναφέρει ότι μεταφορές πίστοσης ε, και οι άμεσες χρεώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 12 και 24 μηνών αντιστοίχως. Θα αντικατασταθούν από το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα βελτιωθεί περαιτέρω. Ο κανονισμός λοιπόν απαιτεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία λαμβάνουν, μάλλον εφαρμοστούν με βάση τον ε, IBAN, τον Διεθνή Κωδικό. τελικά τα ISO 24-22 XML θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες ε, τις μεταφορές πίστος και άμεσες χρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν παρούσα στην ακρόαση της Επιτροπής τη 17η Νοεμβρίου 2010. Πολλά από όσα δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι συζητήθηκαν ε, και σε ύστερο χρόνο, συζητήσαμε από κοινού αφού ε, συλλέξαμε όλες τις προτάσεις. Πάντως ε, δείξαμε ιδιαίτερο ανοιχτό πνεύμα προς όλους τους εμπλεκομένους. Προσπάθησα να συμπεριλάβω όλα τα προβληματικά σημεία και θα ήθελα να σας τα παρουσιάσω πρώτα απ' όλα. Οι ημερομηνίε. Ορισμένοι προτείνουν ότι θα πρέπει να έχει, υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία η οποία θα είναι 24 μήνε μετά από τη θέση ισχύ του κανονισμού. Συμφωνώ με τα ε, στενά χρονικά όρια. Λοιπόν, 24 μήνε θα είναι ε, η πιο μακρά περίοδο που μπορούσα να δεχτώ. Ιανουάριο 2013-2014. Ορισμένοι προτείνουν ότι χρειάζεται να λήξει αυτή η ενδιάμεση περίοδο νωρίτερα. Αν προτείνουν διαφορετικές ημερομηνίε για τους ε, πιστωτές. Δεύτερον, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι διαρωτώνται κατά πόσο είναι σωστό η Κομισιόν να να θέσει με, να προωθήσει πράξεις ε, εξουσιοδότησης ε, για τον τομέα αυτό. Εμείς ε, δεν συμφωνούμε διότι έτσι το πράγμα ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. Ε, η Κομισιόν θα πρέπει να έρθει σε διαβουλεύσεις με τους ε, άμεσα εμπλεκόμενους ε, πριν από την τροποποίηση μη ουσιοδών στοιχείων του κανονισμού. Τρίτον, φαίνεται πως υπάρχει η ανάγκη να εξετάσουμε πώς μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κανονισμός έτσι ώστε οι αλλαγές να μην συμπέσουν. τα τεχνικές απαιτήσει. Ε, αυτό το θέτουν πάρα πολλέ τράπεζε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ρήτρε προστασία του καταναλωτή και που επηρεάζει το βασικό μοντέλο είναι να θεωρώ ότι αυτή η επιλογή που έγινε είναι εσφαλμένη. Αλλά μια που η επιλογή έχει ήδη γίνει τότε οι πελάτες θα πρέπει να τύχουν των απαραίτητων εγγύσεων. Εδώ δεν πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα και άρα οι ρήτρε αυτές θα μπορούσαν να μεταφερθούν από το παράρτημα στον, ε, στον κύριο κανονισμό, στο διαρακτικό. Τώρα, η το θέμα των τελών ή των προμηθειών. Η Κομισιόν προτείνει ότι δεν θα, πρέπει να καταβάλλεται προμήθεια εάν ε, υπάρχει άρνηση πληρωμής, ε, επιστροφή κλπ. Πάντως κάποιες τράπεζες θέλουν να διατηρηθούν οι προμήθειες και το βασικό επιχείρημα είναι ότι σε πολλά υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός με τις άμεσες ε, χρεώσεις ε, οι τράπεζε ζητούν ε, να καταβάλλεται μια προμήθεια. Επειδή εκατοντάδες δισεκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εμπλέκονται σε αυτές τις προμήθειες, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι σημαντικό. Εγώ εξετάζω ακόμα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Εάν υπάρχει γίνονται άμεσες χρεώσεις ε, για τις ε, μεταφορές, τότε θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ανώτατα όρια. Και αυτά θα πρέπει να βαίνουν μειούμενα. Η καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία θέση ισχύ του κανονισμού. Έκτον, υπάρχει και το ζήτημα του γερμανικού ELB. Πολλοί καταναλωτέ ε, ίσως να μην γνωρίζουν ότι χρησιμοποιώντα ε, την κάρτα στο, σε ένα κατάστημα ξεκινούν τον μηχανισμό της ε, άμεσης χρέωσης. Και υπάρχει μια πρόταση τα έτη να μειωθούν σε 3 από 5. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι Γερμανοί συνάδελφοι στην αίθουσα, νομίζω πως το παρόν δεν υπάρχουν. Προκειμένου να μας σχολιάσουν αυτό το γερμανικό πρόβλημα. Και έφοδομον και τελευταίο, Πολλοί επιθυμούν οι μεταφορές πίστοσης να μάλλον να αναφέρεται ότι δεν ε, θα εφαρμοστεί στις ε, μεταφορές. και στις συναλλαγές υψηλής αξίας. Ε, συμφωνώ πως θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική αλλά και ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εφαρμογή του ISO 2021. Οι ενδιαφερόμενοι έθεσαν αρκετές προτάσεις, τροποποίησεις που αφορούν στο άρθρο 2.16 αλλά και σε άλλα σημεία του κανονισμού Να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Κομισιόν για μια η ικανοποιητική συνεργασία η οποία φαντάζομαι πως θα συνεχιστεί και θα έχουμε την ε, έκθεση έτοιμη προς μετάβραση σε ένα μήνα. Θα οργανωθεί ακρόαση με τους ε, ενδιαφερομένους στις 20 Απριλίου στην Επιτροπή ΕΚΟ και θα υπάρχει ένας μήνας για την κατάσταση τροπολογιών. Επίσης οργανώνουμε ένα σεμινάριο του ΣΥΠΑ για τον κανονισμό, το οργανώσαμε μάλλον στις 3 ε, Φεβρουαρίου και ε, είχαν κληθεί όλοι οι εισηγητέ και και κλπ. Ευχαριστώ του συναδέλφους που παρέστησαν. Είχαμε μια ικανοποιητική και καρποφόρα συζήτηση και προσβλέπω το να συζητήσω με τους ε, σκιώδεις συντάκτες ε, το συντομότερο δυνατόν και δει στο Στρασβούργο την προσεχή εβδομάδα. Και τώρα περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας για την μετάπτωση του ΣΕΠΑ και σε κάποια ε, αντιφατικά και προβληματικά σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος είναι εδώ, η Σοφή. το λόγο. Ναι. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη που ήρθα τόσο αργά. Α, προσπαθώ να βρίσκομαι ταυτόχρονα σε διάφορε επιτροπές, παρά που δεν είναι πάντα πολύ επιτυχές. Θα είμαι συντομότατη, γιατί τα περισσότερα μου σχόλια θα τα υποβάλλω όταν έχουμε το έγγραφο μπροστά μα, αλλά από τις πρώτες ανταλλαγές υπόψεων νομίζω ότι ευθυγραμμιζόμαστε στις απόψεις μας. Έχουν δύο θέματα που θα θέλω να θίξω. Το ένα είναι το χρονοδιάγραμμα και οι προθεσμίες. Βέβαια, έχουν αρχίσει οι παρουσιάσεις και πολλοί λένε «Α, όχι, νωρίτερα από το 2014» γιατί τότε υπάρχει φυσικό, φυσιολογική ε, προθεσμία για τις επενδύσεις. Ε, δεν ξεχνίζεται από σήμερα. Ακόμα και αν είχαμε πει 2014, πολλοί οργανισμοί θα ε, δεν θα μπορούσαμε να συμμορφωθούμε την προθεσμία αυτή. Λοιπόν, αν είχαν κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουν στο παρελθόν, ίσως δεν θα χρειαζόταν αυτή η νομοθεσία για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεύτερο θέμα, που δεν είναι απαραίτητο τμήμα του φακέλου, αλλά σχετίζεται, είναι το θέμα των τελών για τις συναλλαγές Είχαμε μια πρώτη ερώτηση προς την Κομισιόν και απάντηση που λέει ότι η Κομισιόν δεν έχει καθησυχαστεί ότι το θέμα αυτών των τελών έχει επιληθεί πλήρως και έγκαιρα. Και ίσως για τις κάρτες το θέμα είναι κάπως ανοιχτό. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η Κομισιόν τι σκέφτεται σήμερα. Γιατί η μέχρι τούδε απάντηση της Κομισιόν δίνει την εντύπωση ότι θα ήθελε να υπάρξει κάποια νομοθεσία στο θέμα αυτό. Όπως είπα θα κάνουμε πιο λεπτομερά σχόλια όταν έχουμε το έγγραφο μπροστά μας και την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών. Πρώτα σε ευχαριστώ. Dirk. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ την εισηγήτρια για ε, την παρουσίαση που μας έκανε. Συμφωνώ μαζί του, ότι οι μεταφορές σε ΕΠΑ ήταν πολύ αργέ μέχρι στιγμής. Πολύ πιο αργέ από ό,τι ελπίζαμε. Όταν πρόκειται η μεταφορά ε, εγχωρίου όγκου κονδυλίων στην ΣΕΠΑ υπάρχει κάποια δράνεια. Επίσης, ο καταργηματισμός ε, οδηγεί στο ότι σήμερα υπάρχουν διάφορα άλλα συστήματα που συνεπάρχουν με τη ΣΕΠΑ και θα εξελιπάρχουν για αρκετό χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι αναποδοτικότητα, επικαλύψεις και λιγότερες δυνατότητες για πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Άρα το αποτέλεσμα είναι κατακαιρματισμό τη εσωτερική αγορά και έλλειψη ανταγωνισμού. Το πιο σημαντικό πολιτικό θέμα τη πρόταση είναι η καταλεκτική ημερομηνία, η προθεσμία όπω λέμε. Από την εμπειρία μου στην ε, Κομισιόν ήταν ότι όταν υπήρχε ορισμένη καταλεκτική ε, ημερομηνία όλοι προχωρούσαν ταχύτατα. Αλλιώς περίμεναν. Το είδαμε αυτό και για την ενέργεια, για τα ταχυδρομεία και για όλα. Δηλαδή όταν υπάρχει καταρκτική ημερομηνία τότε υπάρχει μεγάλη και απότομη πρόοδος γιατί όλοι προετοιμάζονται για την ημερομηνία αυτή. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι κανονισμοί και οι οδηγίε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Θα πρέπει να έχουμε σαφέ χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα όχι πολύ απομακρυσμένο. Να μην αφήσουμε να μα πιώσουν κάποιε ειδικέ ομάδε ε, συμφερόντων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε το γλυκό των δυνατόν να έχουμε μια νέα αγορά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια κατακτική ημερομηνία, μάλλον πιο γρήγορα παρά αργότερα. Thank you very much. Is... Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να λάβει το λόγο, Ζαν Πολ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή, γιατί πάντα μπορούμε να ξαναγράφουμε την ιστορία. Σημαίνει να γνωρίζω κάπως την αρχική οδηγία, γιατί ήμουν εισηγητής. Ε, από ποιο σύστημα λοιπόν ξεκινάμε. Ξεκινάμε από 27 διαφορετικά συστήματα πληρωμών, διατραπεζικών πληρωμών με, πολλές, με διαφορετική αποτελεσματικότητα και ποικίλα κόστη που καθόλου δεν συμβαίνουν τα, τα κόστη αυτά στην αποτελεσματικότητα. Συμβάνουν πολύ, ε, ξέρω πάρα πολύ καλά, μη αποτελεσματικά στήματα εξαιρετικά πανηρά και δεν αναφέρω όνοματα χωρών και το αντίστροφο. Δεν ήταν λοιπόν δυνατό να γίνει εύκολα μια ισχυρή εναρμόνιση και σε πάρα πολλά πεδία ε, αφέθηκε ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής. Αυτό πάλι καθόλου δεν διευκόλυνε τα πράγματα. Επιπροσθέτως, λόγω της δυσκολίας του θέματος και του πολύ μεγάλου κόστους των συναλλαγών, Μπορώ να σα αναφέρω ότι από χώρε που γνωρίζω το πέρασμα στο σύστημα ΣΕΠΑ στοιχίζει πολύ πιο δαπανηρά από το πέρασμα στο ευρώ για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεδομένης λοιπόν αυτή τη πολυπλοκότητα δεν υπήρξε, αν θέλετε, το κουράγιο ή η βούληση ή όλη η ιδέα το να τεθεί μια καταληκτήρια ημερομηνία για, την, για το πέρασμα στο σύστημα αυτό. Τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει μια τέτοια ημερομηνία και επιτέλους τώρα έχουμε ένα καινούριο κείμενο. Μπορούμε λοιπόν, αν θέλετε, να ευχηθούμε και το έχουμε και προσωπικά, να επιταχυνθούν τα πράγματα Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να έχουμε ενάργεια επί του θέματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κρίσιμη μάζα, εφόσον και ενώσο οι δημόσιες διοικήσεις δεν θα έχουν ακόμα εγκαταστήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα ηλεκτρονικών Πληρωμών, δεν θα υπάρχει επαρκής κρίσιμη μάζα. Γι' αυτό λοιπόν και συγχαίρω την εισηγήτρια για την εκπληκτική δουλειά την οποία επιτέλεσε και την αφαρίνω να συνεχίσει με επιμονή και με έντονη την πίστη όπως έχει. Να σας αναφέρω ε, μία λεπτομέρεια που είναι σημαντική. Το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν είχε διευθετηθεί σίγουρα συνεισέφερε στο να καθυστερήσει τις ε, συναλλαγές και θυμάμαι τις όλες τις διαδικασίες και θυμάμαι ότι και εσείς είχατε παρέμβει για να καταρτήσετε, για να καθορίσετε ένα ποσοστό, νομίζω 8 ή κάτι τέτοιο, για μια μεταβατική περίοδο για αυτή την ε, νέα επιτροπή. Ε, για την ε, ΜΥΦ. Οι διάφοροι εμπλεκόμενοι είχαν διάφορες αντιδράσεις. Σε αυτή την επιτροπή λοιπόν των ε, διάστηναλλαγών, την interchange, πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα με σαφήνεια. Αυτό ήταν ε, που επιθυμητό ήταν να μην αναφέρεται σε κανένα κόστος η Επιτροπή αυτή ό,τι αφορά το, το πέρασμα στο σύστημα αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρόκειται, η διαδικασία αυτή είναι εμπορική. Επομένως, οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει να την χάνει κάποια αμοιβή για την δραστηριότητα αυτή, για να καλύπτει το κόστος και να υπάρχει και ένα ε, νόμιμο, αν θέλετε, και λογικό κέρδος. Διαφορετικά καταλείπουμε την οικονομία της αγοράς και περνάμε κάπου αλλού. Ενδεχομένως είναι δυνατόν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε να μετασχηματίσουμε, αν θέλετε, και να περάσουμε το ζήτημα των ηλεκτρονικών πληρωμό να γίνει ένα είδου δημόσια υπηρεσία και δωρεάν. Ξέρω ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο σύστημα σε κάποιε χώρε. Κάποιε χώρε το υιοθέτησαν το σύστημα, κάποιε άλλε το εξάλληψαν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί όπου υπάρχει, αυτή τη στιγμή το κόστο έχει καθοριστεί με φύη τρόπο και έντιμο τρόπο. Εκπληρεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία που δεν είναι και τόσο μισητή. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε να το εξαλείψουμε γιατί θα στοιχήσουν λιγότερο. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου θα πρέπει να πληρωθεί αυτό το κόστο. Γνωρίζω χώρε όπου δεν υπάρχει αυτή η... δεν υπάρχει αυτή η προμήθεια, αν θέλετε, η προμήθεια για τη συναλλαγή, αλλά στοιχίζουν πολύ ψηλότερα, αν θέλετε, ε, σε δανειοδότηση ή αλλού. Γιατί κάπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καλύψουν την υπηρεσία αυτή, να βρουν το κέρδο. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι διαφάνεια, διάβια και λογική. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε αυτή την, ε, αυτή την ε, την ε, προμήθεια διαμεσολάβησης ε, να την, ε, να την βάλουμε, να τη στήσουμε στον τοίχο. Χρειάζεται να υπάρχει. Αυτή η, αφού υπάρχει η προμήθεια αυτή και σε άλλους τομείς, όπως στις πιστοτικές κάρτες ή αλλού. Άρα δεν μπορεί μέσω του κανονισμού αυτού να μην διαθετήσουμε ένα θέμα, το οποίο αν θέλετε είναι και αμφισβητήσιμο και είναι και διεκδικούμενο σε διάφορες δικαιοδοσίες ευρωπαϊκές. Άρα, ίσως δεν θέλω να προκαταλάβω αν θέλετε απόφαση, αν θέλετε δικαστηρίων, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ νωρί η πολύ αργά. Αν θέλετε είναι πολύ νωρί, αν θέλετε πρέπει να περιμένουμε πρωτού παρει προσφυγέ, αλλά ή πολύ αργά πρέπει να το είχαμε διαθετήσει πρωτού υπάρχουν προσφυγέ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πραγματικά εχέφρονε, ρεαλιστέ και ε, προσεκτικοί στην προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ως ε, ε, επίσης ε, επιβιώσας από την οδηγία αυτή που αφορούσε το θέμα των ηλεκτρονικών πληρωμών, έχει διατηρήσει το πάθος που είχες και επέδειξες και το, στις συνομιλίες που είχαν γίνει τότε, στις που είχαν γίνει τότε. Εάν θέλει κανείς άλλος το λόγο, δίνω και πάλι το λόγο στην συγκεντρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Κώστας για την υποστήριξή του και την ενθάρρυνσή του όταν πρωτοανέλαβα την έκθεση αυτή θεώρησα ότι είναι εξαιρετικά τεχνική υφής, ε, αποδείχθηκε όμως ότι υπάρχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα σε όλα αυτά και νομίζω ότι θα το βλέπουμε συνέχεια καθώς προχωράμε. Όπως είπε και η κυρία Σοφμπολτ, δεν θα υπάρχει μια πραγματική ενιαία αγορά αν δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα πληρωμών. Άρα είναι πολιτικός ο στόχος ο οποίος τίθεται. Είναι ένα θέμα προτεραιότητας το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό προσπαθούμε να εισαχθεί και να υπάρξει αυτό το σύστημα ΣΕΠΑ της ε, μιας ενιαίας κοινωτικής αρχής, αν θέλετε, για ηλεκτρονικές πληρωμές. Η κατάσταση στην οποία ε, βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ε, απαράδεκτη δεν μπορεί να συνεχίσει για όλου όσοι έχουν ξεκινήσει και έχουν καταβάλει το κόστο και έχουν κάνει προσπάθεια για να εισάγουν το σύστημα αυτό. Αυτό σημαίνει επιπρόσθετο κόστος για αυτού, γιατί διατηρούν και το παλαιό σύστημα και το καινούριο που έχουν ε, εκπονήσει και εφαρμόσει. Λειτουργούν ε, εκ παραλίλου. Πρέπει κάπω να απλουστεύσουμε τη ζωή εκείνων, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι κινήθηκαν στην αγορά. Ή, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι η ίδια κατάσταση για όλους ε, τους ε, φορείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τα μύφς, αυτά τα τέλη της, ε, της προμήθειας, αν θέλετε, για αυτές τις συναλλαγές, σωστά ε, έδωσε όλες τις παρατηρήσεις ο προλαλής σας, αλλά σίγουρα με τους κοιόδης ηγητές θα καταφέρουν να, να περάσει σωστά το θέμα αυτό. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, πραγματικά προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία, γιατί νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολες, αν θέλετε, πολιτικές ε, γραμμές. Ίσως να είναι, αν θέλετε, εθνικές ε, γραμμές, οι οποίες τίθενται, αλλά όχι σε πολιτικό επίπεδο τόσο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Προθυμένη την αποφυλη των απολογιών είναι 16 Μαΐου. Μαΐου. Θα το εξετάσουμε αρχές Ιουνίου και στις 7 Ιουνίου θα ψηφίσουμε πάνω σε αυτό και 15 Φεβρουαρίου είχε συμφωνηθεί ότι θα υπάρχει μια ακρόση για την ΣΕΠΑ που θα γίνει 13 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα σήμερα είναι οι ψηφοφορίες, αλλά στις 5 παρα 10 έχουν προβληθεί. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα λοιπόν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους παρόντες. Θα πρέπει να επανέλθετε γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 12 μέλη για να ψηφίσουμε. Και μια που είπαμε 5 παρα 10 και ξέρω ότι πολλοί θέλουν να έρθουν, θα αναγκαστούμε να έχουμε μια διακοπή για 20 λεπτά. Παρακαλώ να επανέλθετε όμω. Otherwise you'll have to do it in Strasbourg. θα αναγκαστεί να γίνει αυτό στο Στρασβούργο. Okay, if you could take your seats, then we can proceed. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις πληροφορίες αυτές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Είμαστε αρκετοί, νομίζω δεν χρειάζεται να μετρήσω. Il a dit que je pense qu'on est déjà suffisamment nombreux. Ah oui, Ωραία, παρακαλώ, τοποθετήστε τις κάρτες σας ε, στα μηχανήματα. Να κάνουμε ε, δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, παντήστε τα κουμπάκια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, περιμένετε γιατί διανύμουμε κάποια έγγραφα. Ναι, μα δοκιμάζουμε, δοκιμάζουμε, τεστ, τεστ κάνουμε. Ψηφίστε παρακαλώ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 Okay, if you plug your cards in, do your test vote. Παρακαλώ. Δοκιμάσαμε. 28 μέλη είναι παρόντα, αρκούν και περισσεύουν. Right, everybody got them? Right, well, we'll, we'll, we'll... Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο θέμα προς ψήφιση αφορά τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων. Έχουν διανεμηθεί τα έγγραφα, εντάξει. Ωραία. Συμβαστική πρόταση α. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στο β. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στο συμβαστική πρόταση γ. Συν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται σε τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 12 υπέρ κατά υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου τροπολογία 12 ψήφι κατά αποχές δεκτή τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συνδεσμός Ι. Υπέρ κατά αποχές δεκτός. Συνδεσμός F. Υπέρ κατά αποχές δεκτός. Τροπολογία 17. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία G. Συγγνώμη, G υπέρ κατά αποχές δεκτός. Λοιπόν, θα σφίσουμε τώρα ηλεκτρονικός ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. 28 ψήφισαν, 28 ψήφοι υπέρ. Ομοφωνία. Καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, δεν ακούστηκε το σχόλιο. Και τώρα περνάμε στο σημείο 7 Πρόκειται για την ψηφοφορία των μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Ξεκινάμε με την τροπολογία υπέρχον 13, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά καλύτερα να σε παληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας υπερθύμων 32 ηλεκτρονικός παρακαλώ ψήφισαν άπαντες απορρίφθηκε δίκιο είχα 16 ψήφους κατά 13 υπέρ τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Τροπολογία 33 ε, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές ε, δεκτή. 19 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 34 έχει αποζηθεί. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αν θέλετε μπορούμε να επαληθεύσουμε, είμαι όμως πεπισμένη. Θέλετε να έλεγχο, εντάξει, ψηφίζουμε επί της 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες, όντως απερίφθη. Τροπολογία 35, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 21, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 22, υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. Το 23 υπέρ κατά εποχές δεκτή. Συμβασμός A ψήφι υπέρ κατά εποχές Νομίζω πως έγινε δεκτή, αλλά σε παληθεύσουμε καλού κακού. Ε, παληθέψει επί του συμβασμού Α. Ψήφισαν άπαντες. Έληξε ψηφοφορία. Όντω έγινε δεκτή. Τροπολογία υπερθμών 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβασμός B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή νομίζω αλλά σε επαληθεύσουμε 37 τροπολογία. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. Συγγνώμη, ήταν κάπως συγκεχημένη ψηφοφορία προηγούμενα. Τροπολογία 27 ψηφ Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα περνάμε την τροπολογία 2 σε δύο τμήματα το ξέρετε, το ξέρετε μάλιστα πρώτο τμήμα της τροπολογίας 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 5 υπέρ, κατά, εποχές, δεκτή. 6 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά, 29 παρακαλώ, παραλαμβάνουμε υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβασμός C υπέρ, κατά, αποχές, δεκτός. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Το 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συνεχίστε να ψηφίζετε. 28 ψήφοι υπέρ, 29 ψήφοι υπέρ και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε επί του ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου. Hans Peter Martin, έχεις να προσθέσεις κάτι. Δυστυχώς δεν έχω την κάρτα μου, ψήφισα αποχή. Εντάξει, 29 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 2 αποχές επί του τρομένου επί του τροποποιηθέντος κειμένου και τώρα νομοθετικό ψήφισμα είπε να ψηφίσουμε. Συν μία ψήφος υπέρ και συν μία αποχές. 31 και 2. Λοιπόν, ήταν το αποτέλεσμα.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 Well, we, I think a little bit ahead. Yeah. I think we'll use the extra 10 minutes. The rapporteur is there. Yep. And shadow council. Okay. Leonardo. Okay. I'd like us to. Λοιπόν, θα ήθελα αμέσως να περάσουμε στο σημείο 8. Έχουμε 10 λεπτά πιο νωρί είμαστε από ό,τι ήταν, ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε 10 λεπτά παραπάνω για να συζητήσουμε πάνω στην έκθεση αυτή. Ο εισηγητή και όλοι οι σκιώδε είναι παρόντε. Παρακαλώ, μη συζητάτε κατευθείαν στην αίθουσα, αν θέλετε περάστε έξω. And I'll give the floor to the rapporteur. Και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κάνα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μόλι ήρθα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που όπω συζητήθηκε με τη γραμματεία έχουμε όλε τι μεταφράσει ε, μπροστά μα. Η γερμανική που ήταν ε, το πρώτο κείμενο, η αγγλική που είναι η πιο σημαντική μετάφραση και θα ήθελα καταρχήν να συζητήσω με τους συναδέλφους σήμερα μια που όλοι είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις τροπολογίες δεν θα τις αναφέρω αναλυτικά λόγω τεχνικών ε, προδιαγραφών. Έχουμε 135 τροπολογίες. Α, όχι, 125, διορθώνω. Αλλά... Πραγματοποιήθηκαν αυτά που παρουσιάστηκαν αρχές Φεβρουαρίου. Ε, τα κριτικά θέματα αναφέρονται στην επεξηματική έκθεση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά την πρόταση του κανονισμού της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια καλή πρόταση που αφήνει όμως ανοιχτά κάποια σημεία. Στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή έχουν αποτελματωθεί συζητήσεις. μετά από πέντε συνεδριάσει τη ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούν στα πιο σημαντικά θέματα. Έχω αφήσει ορισμένα σημεία ανοιχτά στην έκθεσή μου για τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή. Το μέσο εφαρμογής καταρχήν στην πρόταση Κομισιόν. Όπως και η προτάση της διάσκεψης κορυφής αναφέρεται στα εξοχρηματιστικά ε, εξοχρηματιστηριακά ναι, παράγωγα. γιατί λέγεται ότι εκείνα που υπάρχουν στα, μέσα στα χρηματιστήρια έχουν ήδη καλυπτεί. Αυτό είναι βέβαια ένα επιχείρημα που θα πρέπει να σκεφτούμε. Από την άλλη μεριά δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλοι ε, συμφωνούν ε, με αυτή την ερμηνεία διεθνώς. Δεύτερο, η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογή, το πιο σημαντικό θέμα, το πιο δύσκολο. Ορισμένοι ζητούν εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Στην Αμερικανική νομοθεσία και είχαμε συνεννοηθεί στην αρχή ότι κατά το δυνατόν θα προσαρμόζαμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην Αμερικανική. Η Αμερικανική λοιπόν προβλέπει εξαιρέσεις για κάποιους τομείς, τράπεζες, μικρές και μεσαίες ε, τράπεζες και τα μιευτήρια... Αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα μια ακρόαση από την Αρμόδια Επιτροπή στις ΕΠΑ, όπου λέγεται ότι θα διακανονίζονται τα παράγωγα αυτά μόνο εάν αφορούν το συγκεκριμένο τομέα. Και όλες οι τράπεζες που έχουν ένα όγκο κάτω από 10 δισεκατομμύρια θα εξαιρούνται γενικά από το πεδίο 10 δισεκατομμύρια δολάρια, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε δις ευρώ, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θα εξαιρούσε πολλές ε, περιφερειακές τράπεζες από την υποχρέωση ε, καθάρισης, θα είχαμε δηλαδή κατά βάση με ένα κανόνα de minimis. Θα έλεγα να περιμένουμε τα αποτελέσματα της ακρόασης αυτής της ΕΠΑ ΕΕ και να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Μετά υπάρχει και μια άλλη εξαίρεση που συζητιέται που αφορά επιχειρήσεις μεσαίες όπου προβλέπεται η θέση ρύθμιση ενός δεκανοσμού de minimis στο ένα δις ετήσιο κύκλο εργασιών. Εκ αυτό αυτός φαίνεται το πολύ ψηλό κατόφλι. Αυτό σημαίνει όμως ότι στην αντίθετη περίπτωση θα εισαγάγαμε υποχρέωση εκαθάρισης για μεγάλες μεσαίας τάξης επιχειρήσεις, παρά μου λογικό, δεν θα ήταν λογικό. Μετά, Υπάρχει μια συζήτηση στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου, προτάση της Γαλλίας, για την κατάργηση του κατοφλίου πληροφόρηση και καθάρισης, όπου λέγεται ότι θα πρέπει μόνο τα ε, παράγωγα να υπάγονται σε υποχρέωση ε, καθάρισης. Βέβαια το πρόβλημα της οριοθέτησης των κερδοσκοπικό και εμείς κερδοσκοπικό είναι πολύ πιο δύσκολο παρά να έχουμε κατόφλι κύκλου εργασιών. Αυτά είναι τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο. Αναφέρθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης για συνταξιωτικά ταμεία, αλλά δεν υπάρχει πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο η ελληνική Κυβέρνηση προτείνει κάποια διαφορετική μέθοδο. Δημόσιες τράπεζες, ενέργεια, ε, ταμεία ακινήτων. Όλα αυτά είναι το μίσους που θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να εξαιρεθούν ή όχι. Μετά υπάρχουν προτάσεις για την ενημέρωση, άρθρο 25 MIFID, όπου υπάρχει ήδη υποχρέωση ενημέρωσης και λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματική υποχρέωση ενημέρωσης. Το κατόφλι ενημέρωσης διαφυσβητείται στο Συμβούλιο και εγώ το διάγραψα. Και η η ομάδα εργασίας αυτή του Συμβουλίου θεωρεί ότι θα μπορούσε επίσης να υπάρχει μία, ε, ένας κανόνας εντεμίνιμης για τις ΜΜΕ. Άλλο σημαντικό σημείο, συνεργασία μεταξύ εθνικών υποπτικών αρχών και ΕΚΑΑΑ όπου λέγεται ότι θα υπάρχει πάρα πολύ ε, πολύπλοκο σύστημα μεταξύ των εποπτές των εθνικών εποπτικών χωρων και ΤΙΑΚΑ και γι' αυτό εγώ ήθελα να το διαγράψω αυτό και να προβλέψω μια ενδυναμωμένη συνεργασία των ε, εποπτικών αρχών και ΑΚΑ Και επίσης α, τοποθέτηση βάση του άρθρου 15 που θα πρέπει να δίνεται στι εθνικέ εποπτικές αρχέ και να υπάρχει και το δικαίωμα δημιουργία και άλλων εθνικών εποπτικών αρχών που θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά του στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μετά, άδειε και των συμβαλωμένων τρίτων χωρών. Αυτό είναι πολύ κεντρικό θέμα. Όπου προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο εύκολη πρόσβαση. Στη δική μου πρόταση προβλέπω εξίσωση των ε, κανονισμών έγκρισης ε, χορήγησης αδείας. Και μόνο σε περίπτωση αμοιβαιότητας θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ή πλήρης ή μερική απαλλαγή από όρους και διαδικασίες της χορήγησης άδειας. Αυτό είναι κάτι που αφορώ εδώ και πολλά χρόνια της είπα. Διαλυγωγικότητα. Και διάγραψα. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, ε, ε, εμφάνισης νέων συστημικών κινδύνων και κάπου ορισμένε προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα βέβαια στη λειτουργικότητα. Υποχρέωση καθάρισης για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλόμενους και τα εξωχρηματιστηρικά παράγωγα που χρησιμοποιούν που δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από μία και μοναδική υπέρβαση του κατοφλίου εκαθαρής, αλλά μόνο σε περίπτωση υπέρβαση του κατοφλίου επί 90 συναπτές ημέρες. Αυτή η ιδέα είναι πιο λογική παρά να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών και να υπάρχει έτσι μια καλύτερη ασφάλεια νομική. Και η, ε, στη συνέχεια θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν μέσα στο χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις εκαθάρισής τους σημαντικότατη αλλαγή αυτή έναντι της πρότασης της Κομισιόν για τις, ε, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλόμενους. Και θα πρέπει μετά από μια ακρόαση να οριστούν τα, τα κατόφλια αργότερα για να ακουστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προτού ε, εδραιωθούν αυτές οι προτάσει στα κατόφλια. Ένα πολύ αφιλεγόμενο θέμα είναι η δρομική ισχύ των υποχρεώσεων. Η καθάριση συμβάσεων εξοξωματιστικών παραγωγών που έχουν ήδη αναφερθεί, το λεγόμενο backloading. Εγώ για νομικούς λόγου, θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω της εκ των υστέρων ασφάλειας. η αναδρομική υποχρέωση δήλωσης είναι διαφορετικό. Είναι δυνατόν να ισχύει η αναδρομική υποχρέωση αναφοράς ανάλογα με την κατηγορία παραγόγων, την αναπομένουσα λικτότητα και τις τεχνικές προϋποθέσεις. Και θα πρέπει να υπάρχει και ταξινόμηση ανάμεσα, ε, ανάλογα με ταξινόμηση των παραγόγων και να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τα οικονομικά στοιχεία. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που προτείνονται και θα με ενδιαφέρε, χωρίς να επαναλάβω όλες τις τροπολογίες, ποια είναι η άποψη των συναδέλφων από αυτών. Προτίθεμαι μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων εδώ στην Επιτροπή, να επιδιώξω ευρεία συνένεση, η οποία θα αντικατοπτρίζει το στόχο της, ε, του κανονισμού να διακανονίσει δηλαδή τα παράγωγα αυτά χωρίς να δημιουργήσει νέα συμπληρωματικά οικονομικά εμπόδια που θα οδηγήσουν σε δυσάρεστο κόστος και σε σημαντική μείωση της αγοράς. Τούτον να σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συνενετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Λεωνάρδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε ευκαιρία να εξετάσουμε τις τροπολογίες και διάφορες, γλωσσικές εκδοχές και έχω την εντύπωση πως ε, αυτή είναι μια πρώτη ευκαιρία για να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων επί της ουσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα μου θα καταρτήσει και θα παρουσιάσει εντός ε, της προθεσμίας ε, της τροπολογίας της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις ε, του εισηγητή κ. Λάγκεν, θα ήθελα να τονίσω κάποια συμφωνία επί των οποίων συμφωνούμε και κάποια άλλα που κατά την άποψή μου απαιτούν ε, μια περαιτέρω ευάθυνση ή που προκαλούν σε εμά και ιδιαίτερα σε μένα ως και ηγητή ορισμένους προβληματισμούς και επιφυλάξεις. Όπως ήδη δήλωσα την προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων συμφωνώ με, την, ε, με το ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού να αφορά αποκλειστικά τα έξω παράγωγα και έτσι μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα δήλωσε ο κύριος Λάγκεν. Έχω κάποιους προβληματισμούς και ανησυχίες επίσης επί του σημείου που αφορά τις εξαιρέσεις, τις παρεκκλήσεις, διότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ε, περιορισμό, έναν μετριασμό θα λέγαμε της δέσμευσης που ε, είχαν ε, αναλάβει και στο πλαίσιο του G20. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να επιλέξουμε κάποιοι και να καθορίσουμε κάποιες αρχές με βάση ορισμών που κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακόμα σαφείς, όπως το ζήτημα του περιορισμού μόνο σε προϊόντα που έχουν συστημική σημασία. Να πω επίσης ότι δεν κατάλαβα καλά και θα ήθελα μια εξήγηση περί αυτού το σημείο που αφορά στις εξαιρέσεις ε, ε, με βάση τον ε, κύκλο εργασιών μιας τράπεζας. Ο κύριος Λάγκεν αναφέρθηκε στις ακροάσεις που διεξάγονται και στην Αμερική αλλά και ακόμα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω πως ε, το ζήτημα εδώ είναι να προσδιορίσουμε ποιο είναι το κατόφλι το οποίο χρειάζεται να λάβουμε υπόψη. Ε, να πω επίσης με τα σημεία στα οποία διαφωνώ, ε, συμφωνώ το ζήτημα των ε, αδειών η κατάργηση του σημείου που αφορά την ε, διαλειτουργικότητα αλλά και το ζήτημα του backloading. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, επί της ουσίας σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε κάποιες ε, τροπολογίες. Το πρώτο ερώτημα που θέτω αφορά στην τροπολογία υπερθμών 51. Διαρωτώ με λοιπόν εάν όντως θα ήταν χρήσιμο να διαγραφεί το κείμενο της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον αναφορά της υπέρβασης του κατοφλίου σύμφωνα με την παραγραφό 3α. Κατανοώ την πρόθεση του τροπολογίας και τον λόγο υπαρξής της, ότι δηλαδή θέλουμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό κόστος, αλλά διερωτώμε κατά πόσον η διαγραφή αυτού του τμήματος ε, του άρθρου 7 του κανονισμού που προτείνει η Κομισιόν δεν θα προκαλέσει κάποια προβλήματα από πλευρά διαδικασία και ως εκ τούτου να αποδυναμώσει, την ισορροπία της, ε, του όλου διατάγματος ε, τώρα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 53 ε, και 54 ειδικά συγγνώμη τροπολογία 53 και εδώ κατανοώ τη σημασία που βρίσκεται στην βάση αυτής της ε, τροπολογίας ε, που αφορά στην ε, υπέρβαση σύντομη διάρκεια των κατοφλίων αντιστάθμισης, αλλά οι 90 ημέρες διερωτώ με αν θα μπορούσε να θεωρηθεί μια σύντομη χρονική περίοδος. Κατά την άποψή μου πρόκειται για μια περίοδο αρκετά ουσιαστική, αρκετά σημαντική και μακροχρόνια θα έλεγα. Τώρα και μια περιττέρου παρατήρηση σχετικά με τροπολογία υπαριθμών 64. Συμφωνώ με την αρχή της ε, ε, περιουσιακής βάσης η οποία θα πρέπει να είναι πιο σταθερή πιο ισχυρή και ως εκ τούτου η ε, αύξηση του αρχικού κεφαλαίου πέραν ε, των προβλεπόμενων από την Κομισιόν δηλαδή 5 εκατομμύρια ευρώ διαρωτώ με εάν ε, το να ανεβάσουμε στα 10 εκατομμύρια το ποσό επαρκεί ή δεν απαιτείται να πάμε ακόμα πιο μακριά, να κάνουμε ένα ακόμα βήμα αυξάνοντας ε, περαιτέρω το αρχικό κεφάλαιο και να πω δύο Λάγκεν ότι στην, ε, εκτιμώντα το σημείο Δέλτα όπου γίνεται αναφορά στην ε, αδειοδότηση των ανισφαλωμένων κλπ. Μιλάμε για αρχικό μόνιμο κεφάλαιο της τάξης τουλάχιστον 5 εκατομμύριων ευρώ, αλλά φαντάζομαι πως ο κύριος Λάγκεν, σύμφωνα με τα όσα πρότεινε ως εισηγητής στις τροπολογίες, επιθυμεί να τροποποιήσει αυτό το ποσό. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις παρατηρήσεις ε, γενικού χαρακτήρα αλλά και ιδιαίτερου χαρακτήρα που θα ήθελα να κάνω και καταλήγω λέγοντας ε, ότι για μένα αυτό που είναι θεμελιώδη ζήτημα και πιο λεπτό είναι το σημείο που αφορά το ζήτημα των εξαιρέσεων, των παρεκκλήσεων, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το σημείο το οποίο αν δεν ε, εξετάσουν με τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό μπορούν ε, να ανοιχθούν οι διάφορες ε, θύρες θα έλεγα που από που τελικά θα διεισδύσουν κάποια στοιχεία που θα επηρεάσουν το όλο νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά σημείωνα ακόμα όντας ε, σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα φιλελευθερών. Θα υποβάλλω τη σχετική, καταρχάς θα πιο την αντίδρασή μου στον ε, εισηγητή. Καταρχάς να ευχαριστήσω για το ότι επανέλαβε και επανέφερε κάποιες από τις παρατηρήσεις που είχα υποβάλει εγώ στη γνωμοδότησή μου από την Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων. Και ξέρω ότι είναι χρήσιμο. Ε, ας διατρέξουμε τα ανοιχτά ζητήματα Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, με ενδιαφέρει πραγματικά να υπάρχει ισότιμο παιχνίδι. Σε κάποιο βαθμό, λοιπόν, υποστηρίζω την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα. Και ιδιαίτερα νομίζω ότι εάν θέλουμε να έχουμε μια συνολική επισκόπηση των θέσεων και θέλουμε να τις δούμε ομαδοποιημένα στην, ε, ε, στις, ε, στα αποθετήρια, νομίζω ότι όλα γιατί θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικές, ε, στα σχετικά αποθετήρια. Γιατί ήδη είναι σε ηλεκτρονική μορφή τα αποθετήρια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τα αρχεία εγγραφών, τα αποθετήρια, νομίζω ότι η Επιτροπή έχει απόλυτα δίκιο ότι θα πρέπει να ισχύει τα όσα διέπουν τα σχετικά αρχεία καταγραφής, ε, όλα ανεξαιρέτως τα παράογα. Ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη σκέψη, ίσως μπορούν να το γνωστοποιήσουν. Τώρα, εάν η ακαθάριση ε, στα χρηματιστήρια ή αν θέλετε οτιδήποτε είναι και λειτουργεί ως χρηματιστήριο, γιατί ξέρω ότι τώρα μπαίνουμε λίγο σε κρίζα ζώνη, με τις ε, διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν. Εάν δεν είναι η εκαθάριση όσο ισχυρή, αν θέλετε, και στεναρή όπως πρέπει να είναι, πρέπει να την κάνουμε εξίσου όπως θα είναι για τα εξοχρηματιστηριακά παράγοντα. Δηλαδή οτιδήποτε ισότιμο, αν θέλετε, σίγουρα δεν χρειάζεται να υπάρχει διπλίως και επικάλυψη κανονισμών, αλλά πάντως θα πρέπει ίσως να υπάρχει κάποια γλώσσα που θα μας επιτρέψει να καλύπτουμε, διατύπωση που θα καλύψουμε, αν θέλετε, κομματάκια που ενδεχομένω μας λείπουν. Τώρα, στις εξαιρεσει για τους αντίστοιχους λόγους θα έλεγα, Νομίζω ότι από πλευρά ε, και πάλι των αποθετηρίων, των αρχείων καταγραφή, δηλαδή, πάλι θα πρέπει να δούμε, γιατί συστημικό κίνδυνο υπάρχει. δεν είναι στου θεσμού ο συστημικό κίνδυνο, είναι στο σύστημα. Πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε σε το συστημικό κίνδυνο, σε σχετικά ε, ιδρύματα, οργανισμούς αν θέλετε, που εμπλέκονται στο σύστημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μικρομεσαίοι οργανισμοί που λειτουργούν με αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν συγκεκριμένους δείκτες όπως το που ενδεχομένως έγκυται και δομείται συστημικός κίνδυνος δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ότι συστημικός κίνδυνος υπάρχει μόνο σε συστημικά πολύ μεγάλους οργανισμούς. Μπορεί να είναι διαφορετικός, αλλά μπορεί να τύχει αντίστοιχη διαχείριση. Με προβληματίζει λοιπόν η εξαίρεση και η παρέκκληση. Εγώ δηλαδή πραγματικά δεν θα βάζα εδώ πέρα, δεν θα ήθελα να, να υπάρξει κάποια εξαίρεση ή παρέκκληση σε ό,τι αφορά τα αρχεία καταγραφή των συναλλαγών. Βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει στο αποτέλεσμα της ακρόασης. Αλλά, για παράδειγμα, οι περιφερειακές τράπεζες, οι οποίοι λειτουργούν με αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντήλα, μοντέλα, θα έπρεπε να μην εξαιρούνται. Είδαμε να υπάρχει συστημικό κίνδυνος στην ε, ε, Ισπανική τράπεζα. Γιατί δεν θα υπάρχει το ίδιο κίνδυνο και με τα, χρηματο... και με τα ε, παράγωγα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατόφλι, προσπαθώντα να καθορίσουμε τι είναι κερδοσκοπικό, αν θέλετε, όριο, θα είναι όντω δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσον το θέμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τον όλο προβληματισμό με τα σεξουαλικά ταμεία. Πρέπει και πάλι να δούμε τι θα κάνουμε. Θα επιτρέψουμε κάποιο επίπεδο ε, εξοχρηματιστηριακών παραγόγων να συνεχίσουν να λειτουργούν. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει αντίστοιχα, αν θέλετε, ισχυρό και υγιές ε, σύστημα για δι... εκαθάρισης διμερών συναλλαγών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τα συγκριτικά ταμεία και για άλλους σχετικούς θεσμούς. Η εναλλακτική, αν δεν λειτουργήσει αυτό, θα είναι ίσως να δούμε τις, όλες τις θετήσεις που υπάρχουν για τις ε, κινητές αξίες ε, και τα χέγγια. Γιατί γενικά, εάν όλα αυτά προκαλούν μεγαλύτερες δαπάνες στα ασφαλιστικά ταμεία, τελικά δεν εξυπηρετούμε τον πολίτη. Σύμφωνο πιθανότατη ότι θα πρέπει να, ε, να δούμε και να, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει πληροφόρηση να, έχουμε, να ευθυγραμμιστούμε με αυτά που προβλέπονται από την MIFID. Τώρα, το θέμα του πού εφαρμόζεται αυτό, ίσως θα πρέπει να το δούμε ε, ευρύτερα, ίσως να είναι λίγο λιγότερο σε μικρότερα κράτη-μέλη. Αλλά εγώ νομίζω ότι πάντα θεωρούσα ότι θα έπρεπε ε, να υπάρχει πάντα και να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Επιτήρησης ε, ίσως είναι και λιγότερο και πιο φθηνό αν θέλετε. Σε περισσότερες περιπτώσει, όλες οι κεντρικές τράπεζες θα είναι οι εθνικοί θεματοφύλακες των όλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Άρα ενδεχομένως θα είναι μια πολύ δεξιοτεχνική κίνηση αν θέλετε να παραπέμψουμε όλη την επιτήρηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε και την αμεβαιότητα, δεν είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε στο δικό μα ιστορικό κανονισμό κάτι το οποίο συμβαίνει αλλού και που να μην θέλουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταστεί σαφέ ότι πρέπει να το κάνουμε με βάση των ε, προτύπων ισοδυναμία, ε, όχι απόλυτη ομοιότητα και ισότητα. Θα ήθελα λοιπόν να επανεξετάσουμε λίγο εδώ τη διατύπωση. Τώρα, για κάποιες τύπους θα μπορούσαμε να έχουμε διαλειτουργικότητα, έτσι όπως το έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μην λέμε ότι είναι συστημικός θέλω το κίνδυνο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό σημείο. Όπου μπορούμε λοιπόν με ασφάλεια να έχουμε διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να την εισάγουμε, ενώ είναι λίγο πιο πολύπλοκο το ζήτημα και, και το αποδέχομαι σε κάποια άλλα πεδία, όπου ίσως εκεί θα πρέπει να το αφήσουμε προς το παρόν. Αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θέλουμε να επανέλθουμε. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ του ποιο είναι κερδοσκοπικό και ποιο μη κερδοσκοπικό σε μη χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να νομίζω να έχουμε το ίδιο σκεπτικό με αυτό που είχα εγώ, όπω το εξετάσαμε στην Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων. Γιατί σε ό,τι αφορά τις ε, παρεκκλήσεις που προσφέρονται, που δίνονται στις ε, μεγάλες εταιρείες, ε, ίσως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε στα πλαίσια των ελέγχων που γίνονται, των οικονομικών καταστάσεων και απολογισμών. Τώρα, σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτέ τι εξαιρέσει, μπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηρή η διαδικασία. Όταν ρώτησα, δεν θέλουμε να έχουμε μια διασταύρωση, αν θέλετε, με κάθε συναλλαγή για κάθε παράγωγο ένα προ ένα. Θα πρέπει να είναι δυνατόν όμως με τον ε, ορκωτό λογιστικό έλεγχο να δούμε κατά πόσον ε, λειτουργεί, αν θέλετε, το όλο σύστημα με την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τελείως διαφορετικής κλίμακας, διαφορετικού εύρους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να παίξουμε λίγο με τη διατύπωση του αντικειμενικά μετρήσιμου. Συμφωνώ τώρα σε ό,τι αφορά το αναδρομικό. Νομίζω ότι αυτό το backloading, δηλαδή η καθάριση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγόγων που έχουν ήδη συναυθεί ηλεκτρονικά, είναι όντως πολύ καλή ιδέα και είμαι υπέρ αυτού. νομικά βέβαια παρουσιάζει πρόβλημα. Εάν έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις, θα πρέπει αναδρομικά να ζητήσουμε δώσιμο μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους πιθανόν θα πρέπει, ίσως θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα, να δούμε εάν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα παγκινδυνευμένη και δύσκολη τάξη περιουσιακών στοιχείων, αν θέλετε, περιουσιακών στοιχείων, ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχει διατύπωση αυτή τη στιγμή, δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι με αυτά καλύπτουμε τα περισσότερα από τα σημεία στα οποία θέλετε κάποια απάντηση. Προφανώς υπάρχουν και πολύ περισσότερα. Θα δω αν μπορούμε να τα συζητήσουμε κάτι κατηδίαν αν θέλετε ή να βάλουμε και κανένα δυο ακόμα τροπολογίες. Αυτά. Τώρα, επόμενος που ζήτησε το λόγο, ο Πασκάλ. Εγώ θα είμαι λίγο πιο σύντομος από τη σκιώδη συγγήτρια, γιατί δεν είχα πάρα πολύ χρόνο να μελετήσω την έκθεση και μάλιστα πρέπει να τη μελετήσω τα αγγλικά. Θα είμαι πιο σύντομος λοιπόν και θα έχουμε προφανώς την ε, ευκαιρία να τη συζητήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κατά την κατάσταση τροπολογιών. Το πρώτο στοιχείο επί το οποίο θέλω να επιμείνω αφορά στις εξαιρέσεις τόσο σε ό,τι αφορά τις ε, οικονομίες, τις εταιρείε ε, ε, αν θέλετε, τη εφαρμογή, Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις εταιρείε πραγματικής οικονομίας, και εκεί μπορούμε να έχουμε κάποιες εξαιρέσεις, τώρα σε ό,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς ε, οργανισμούς, δεν βλέπω γιατί πρέπει να ανακατευτούμε εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν κάποια αιτήματα, ξέρεις, αν θέλετε, που έρχονται παντού. Και θα βρεθούμε τελικά να έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος ο οποίος θα είναι σαν δίχτυ, διάτριτο παντού, δεν θα υπάρχει συνέπεια. Άρα θα πρέπει να έχουμε όσο να δω τις λιγότερες εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογή για όσους δεν άπτονται, αν θέλετε, ε, για όσους δεν είναι οργανισμοί της πραγματικής οικονομίας εντός εισαγωγικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά του όλου ε, κολεγίου, αν θέλετε, της, ε, της ΕΑΚΑ, τι θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχει ε, κανονιστικός ανταγωνισμός μεταξύ των ε, διαφόρων ε, διαφόρων ε, αδειών κεντρικών αντισυμβαλωμένων σε ό,τι αφορά αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου. Το ιδανικό θα ήταν, να θέλετε, να έχουμε έναν ενιαίο ε, κανονισμό για από την ΑΚΑ, από όλου. Δηλαδή, αν έχουμε ενιαίου κανόνε, μπορούμε να διαχειριστούμε τον συστημικό κίνδυνο. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, τότε το, το, το κόστος από όλο αυτό το σύστημα διαφορετικών κολεγίων, αν θέλετε, διαφορετικών αδειών, που θέλαν ακριβώς να συγκεράσουν αφενός με την εποπτική αρχή κάθε χώρας και αφετέρου την, ε, το θεματοφύλακα, την εποπτική αρχή των τραπεζών που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις άδειες και που ενδεχομένως έχουν έδρα σε άλλη χώρα από εκεί που βρίσκεται ο αρχικός ε, αντισυμβαλόμενος, κεντρικός αντισυμβαλόμενος. Άρα το κολέγιο αυτό, τα κολέγια αυτά που δημιουργούνται έχουν κάποιο νόημα. Θα ήθελα όμως να δούμε, ε, νομίζω ότι αν ε, αλλάξει αυτή η διατύπωση, δίνουμε υπερβολική ισχύ στην Εθνική Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών, ε, οπότε ξαναβάζουμε πάλι και ξανακινητοποιούμε τα ίδια γρανάζια αν θέλετε, όπου θα πρέπει να έχουμε προσφυγή στο τέλος σε έναν εξωτερικό τελικό διαιτητή, γιατί θα υπάρχει πάλι ανταγωνισμός κανονιστικός μεταξύ των διαφορετικών εποπτικών αρχών. Αναφέρθηκαν, αν θέλετε, οι ανισορροπίες ε, μεταξύ των διαφορετικών χωρών, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα επίπεδο ανταγωνισμού, το οποίο δεν ε, πραγματεύεται παρκώς η έκθεση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα, κατ' επανάληψη τονίστηκε από τις ε, διάφορες πολιτικές. Σωστά πηγαίνουμε, είναι σωστό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση εκαθάρισης, τον κανόνα των 90 ημερών, Νομίζω το καλύτερο είναι να επινοήσουμε, αν θέλετε, μια περίοδο, όχι μια καταληκτήρια ημερομηνία, για να Έχουμε, δηλαδή πρέπει να, να τελειοποιηθεί, αν θέλετε, να, πολύ περισσότερο για τύπωση τη αρχική πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά οι 90 μέρε νομίζω είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντως το ότι θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο ε, χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των ε, ε, καθαρίσεων αυτών θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Τελευταίο σημείο, σε ό,τι αφορά την υποβολή αναφορά, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην υπάρχει κανένα κατόφλι σε ό,τι αφορά τις αναφορές των συναλλαγών και ο νομοθέτης, η εποπτική αρχή, συγγνώμη, να έχει ε, συνολική εποπτεία, απόλυτα διαυγή της αγοράς. Γιατί όταν υπάρχουν διαφορετικά κατόφλια και διαφορετικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα εχέγγυα, ε, τα collateral, δηλαδή και τις διάφορες δραστηριότητε κινητών αξιών, είναι λογικό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνολική εποπτεία τις εποπτικές αρχές. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτά γνωρίζοντα ότι εν γέννη συμμερίζομαι τις ε, προτάσεις και υποδείξεις που έκανε η ομάδα του Σιελστών, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες όταν θα βρεθούμε για την ε, συνέχεια της συζήτησης επί της εκθέσεως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λάγκε. και πάρα πολύ καλά σε ένα πολύ πολύπλοκο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά. Προχώρησε πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία μας έδωσε το έγγραφο αυτό. Πολύ λίγες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για τις περισσότερε συμφωνώ μαζί του όσον αφορά το backloading παραδείγματο χάρη όπως ορίζεται και η αναδρομική εφαρμογή των ε, νομοθετικών πράξεων είναι προβληματική. Όσον αφορά λοιπόν την εκαθάριση, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή ότι αυτό το backloading είναι και περιττό και άδικο. Από την άλλη μεριά συμφωνώ ότι θα μπορεί εκ των υστέρων να υπάρχει υποχρέωση αναφοράς. Αυτό γίνεται. Και για όλους τους ε, τομείς νομίζω. Και θα πρέπει να γίνεται γι' αυτό. Ίσως έχουν συμπληρωματική δουλειά να κάνουν εξ αυτού, αλλά νομίζω θα πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος του συστήματος. Εγώ θα ήθελα να ε, αναφερθώ στο θέμα των ε, επενδυτών, το θέμα ανησυχώ όταν αφορόμαστε στην διαχωρισμό, στην προστασία των ε, επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων. Το θέμα είναι όμως ότι έχουν συζητηθεί διαμακρών, ιδίως μετά το Μέιτοφ, έχει, υπάρχει μια μετατροπή της βασικής προστασίας που προσφέρεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο επιλεκτικοί, προστατεύουμε πολύ καλά τους επενδυτές μας από ό,τι το κάνουν στη ΣΥΠΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μας επιδράσει τόσο πολύ το τι κάνει η Αμερική για το θέμα της προστασίας των περιουσιακών αυτών στοιχείων, γιατί εμείς έχουμε έτσι και υψηλότερα κατόφλια προστασίας. Αυτά τα θέματα των επενδυτών θα πρέπει να είναι λοιπόν πάρα πολύ ψηλά στην, ε, στο κατάλογο των θεμάτων που εξετάζουμε. Και μετά. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη επιλογή. Δηλαδή, εάν οι επενδυτέ χρειάζεται να πληρώσουν περισσότερο για περισσότερη προστασία, γιατί να πούμε όχι. Επίσης, όσον αφορά το θέμα των ε, λεγόμενων υγρών ε, στοιχείων, ασφαλιστικών στοιχείων, collateral. Δεν ξέρω κατά πόσο διαφορετικές μορφές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πλαίσια των διακυπάσεων. Και κατά λίγο στο συμπέρασμα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα συνταξιδοτικά ταμεία που είναι πάρα πολύ ασφαλή ταμεία με πολύ σταθερές ε, στρατηγικές θα πρέπει πραγματικά να εξαιρεθούν. Ίσως αυτή ήταν η μόνη λύση, γιατί αυτή τη στιγμή αν ζητούν ε, να εφαρμοστούν, να εφαρμοστούν συστήματα για κολάτερα, για ασφαλιστικά στοιχεία, δεν υπάρχει κανένα μηχανισμός, από όσο κατάλαβα εγώ, που οι διαγωνισμοί αυτοί μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την ποιότητα των πιστώσεων. Μάλλον ανάλογα με το προϊόν που είναι το αντικείμενο της ε, συναλλαγής. Στα εξωτερικά ταμεία λοιπόν δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι ενέχονται ένα κίνδυνο για το σύστημα και θα πρέπει να τύχουν τις ίδιες μεταχειρήσεις όπως εκείνα που ενέχονται το κίνδυνο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην πληγούν οι οι συνταξιούχοι μας. Μετά, για διαλειτουργικότητα. Έχω κάποια προβλήματα με τη διαλειτουργικότητα και αναρωτιέμαι γιατί κάτι τέτοιο είναι ωφέλιμο ή γιατί μπορεί να είναι προβληματικό για τα μοντέλα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Και τελικά συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι το να υπάρχει ανταγωνιστική αγορά καθάρισης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ΜΥΦΙΤ να μην χαθούν καθοδόν. Και αυτό που ανησυχεί δεν είναι η διαλειτουργικότητα αυτή καθε αυτή, αλλά η ανάγκη να υπάρχουν δικαιώματα πρόσβασης για να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον καθάρισης. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο θεωρεί ότι ίσως έχει, έχουμε περάσει διαφορετικό ταμπλό που παίζουμε. Γιατί τελικά το 90% των συναλλαγών χρηματιστηριακών ε, συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνονται μέσα στα πλαίσια αυτών των διατάξεων και δεν ξέρω και ποιο θα είναι το, το μέλλον, δηλαδή ποιες αγορές θα γίνουν, ποιες συγχωνεύσεις ομίλων θα γίνονται και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο όπως υπάρχει μέσα στα πλαίσια του MIFID. Όλο αυτό που ζητάμε για τα κατόφλια και την μη χρηματοπιστωτική κάλυψη ε, πιστεύω ότι έτσι προσπαθούμε να μην υπάγονται οι συναλλαγές των επιχειρήσεων στην, στην διάταξη αυτή της εκαθάρισης. Γιατί δεν πρόκειται για ε, συναλλαγή, αλλά πρόκειται για ασφάλιση των εταιριών. Και δεν θα πρέπει νομίζω να υπάγονται στην εγκαθάριση. Κατ' ουσία υπάρχει σημαντική διαφορά. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε μία λειτουργικότητα ταμείου και όχι συναλλαγής. Ακόμα και αυτοί που χρησιμοποιούν το AS39 πρέπει να αιτιολογήσουν στους ε, ορκωτούς τους λογιστές περί τίνους πρόκειται. Τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις δυνατότητες που φαίνονται εδώ για την περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ολισκιώδεις. Κοέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον συνάδελφο Λάγκ που παρουσίασε μια έκθεση η οποία θεωρώ πως αποτελεί μια εξαιρετική εργασία. που προχωράει προς την επίτευξη του επιθυμητού στόχου, δηλαδή της μείωσης ε, του κινδύνου και την αύξηση της διαφάνειας ε, στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Αυτές οι προσπάθειες ε, πραγματικά γίνονται και από τις δύο πλευρές του ωκεανού, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Πολιτείες με τον νόμο Frank Dodd Act θα ήθελα να πω ότι τα παράγωγα στη σημερινή οικονομία επιθυμούν να πετύχουν ποικίλου στόχους και μέσω των τραπεζών διακανονισμού επιθυμούν να πετύχουν τον στόχο τους. Ο εισηγητής ήδη έκανε κάποιες προτάσεις βελτιωτικές της ε, πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, εξαιρέσεις. Να ήθελα να τονίσω επίσης τον σημασία του ρόλου που μπορεί να δραματίσει ΕΣΜΑ και πρόκειται για ένα ρόλο ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί κάλλιστα με τα προτινόμενα. Θα ήθελα να τονίσω επίσης πως ε, η κατάσταση των ε, ασφαλιστικών ταμείων ε, που εμπίπτουν στην οδηγία IRP. Πρόκειται για έναν ορισμό ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, ο οποίος ορίζει προϋποθέσεις ιδιαίτερα σαφείς. Γνωρίζω το Ολλανδικό μοντέλο όπου τα ασφαλιστικά ταμεία υπόκεινται σε κάποιες ε, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις ιδιαίτερα υψηλές προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθούν τις ε, πληρωμές, τις καταβολές ε, σε οποιαδήποτε στιγμή. Και προβλέπονται πάρα πολλέ δικλείδε ασφαλεία. Τώρα, αν κάνουμε την ε, συσχετισμό με τα όσα ισχύουν από την άλλη του Ατλαντικού, στι ΗΠΑ, διαπιστώνουμε ότι αυτού του είδου τα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον υπάρχουν σε πολύ μικρότερο βαθμό από στο παρελθόν. Και θεωρώ ότι είναι πράγματι κρίμα αυτού του είδους η αποταμίευση εν ώψη της συνταξιοδότησης που αποτελεί ένα είδος ασφάλειας για τους πολίτες μας να ε, ζημιώνεται. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια λύση, υπενθυμίζοντα πω η διαφάνεια σχετικά με το εμπόριο των παραγωγών είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά φυσικά μπορούμε να αξιολογήσουμε και την δυνατότητα να δεχτούμε δραστηριότητες ε, εγγύησης των ε, εναλλακτικών collaterals. Και καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο πιο σαφείς ε, και πιο ευρύς τους ρόλους των αρχών εποπτείας δεν είναι μόνο η ΟΠΑ αλλά και η ΕΑΚΑ που μπορούν να διαρματίσουν αυτόν τον ρόλο. και να ζητήσουν περισσότερες, ε, περισσότερα χέγγια για αυτού του ίδιου τις δραστηριότητες. Να θυμίσω ότι τα χρήματα των πολιτών μας, χρήματα τα οποία αποταμίευσαν ε, για τη σύνταξή τους από 1,5 δις έως 2,5 δις ε, στις κατοχώρες, Αυτό το κονδύλια λοιπόν θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται με τρόπο λελογισμένο. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος που να επιθυμεί να λάβει το λόγο. Η Κομισιόν. Πάτρικ, έχεις να πεις κάτι. Σύντομα, Πρόεδρε. Πρώτα, σχετικά με το τι θα πρέπει να καθαρίζεται. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ζητιέται στο Συμβούλιο, ότι θα χρειάζεται να επεκταθεί σε όλα τα παράγωγα και όχι μόνο στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Και αυτό για πολλούς λόγους. Αν περιορίσετε μόνο στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τότε το Κοινοβούλιο θα περιορίσει τον ε, πεδίο εφαρμογή στην πράξη, διότι στην αναθεώρηση της ΝΕΦΙΝΤ θα ζητήσουμε κάποιες ε, εγγυήσεις δεν ε, θα απομείνει και πάρα πολλά ω τούτου για να καλύπτονται από αυτήν την νομοθεσία, από αυτή την οδηγία. Και ενδεχομένως να μην χρειάζεται να διεξαχθεί ούτε καν συζήτηση όπως ακούστηκε μπορεί να αποτελέσει ένα κενό σημασίας νομοθέτημα, κενό ουσίας. Εξετάσαμε τα νομικά, νομικές πτυχές με τους νομικούς παίοντες στην Κομισιόν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν και οι ΗΠΑ το Frank Dodd, να μην ε, εφαρμοστεί το backload, και αν κάτι θα πρέπει να καθαριστεί, αυτό θα πρέπει να ε, αποφασιστεί αργότερα. Όχι backloading λοιπόν, αλλά να διαβεβαιωθούμε ότι όταν, εφαρμοσ... όταν αποφασιστεί αυτή η οδηγία θα έχει ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή. Μας υπόθηκε ότι αυτό είναι δυνατόν και ένα άλλο σχόλιο αφορά τις εξαιρέσεις, τις παρεκκλήσεις. Τι θα πρέπει να εξαιρείται. Ε, η αρχική συζήτηση ήταν ε, πολύ σαφή, Θέλουμε μια ισχυρή νομοθεσία και τώρα φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, ισχυρή νομοθεσία μεν, αλλά όχι στην, ε, στα του οίκου μου. Λοιπόν, ασχοληθή, συζήτησαμε το ζήτημα με τις εποπτικές αρχές και η αναφορά που γίνεται στα 10 δις δεν ε, τους βρίσκει σύμφωνους. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μόνο μία εξαίρεση και η επιχείρηση αυτή έχει το 90% της δραστηριοτήτων μόνο σε έναν τομέα. Το θέμα τώρα των ασφαλιστικών ταμείων. Συμφωνώ με, με τα μέλη της Επιτροπής. Υπάρχει πρόβλημα, χρειάζεται να επιληθεί τάχιστα. Το διμερές καθάριση δεν αποτελεί εκαθάριση, μόνο ότι ο όρος είναι ο αυτός. Δεν είναι αρκετά στεναρός Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει αναστabiliτος ορισμός των collateral, χωρίς όμως να επηρεάσουν ε, τον ε, CCP. Τώρα ακούστηκαν και κάποια άλλα επιχειρήματα τα οποία χρειάζεται να εξεταστούν περαιτέρω. Στην ακρόαση δεν είναι απαραίτητο. Το άρθρο 15 της ε, ΕΑΚΑ προβλέπει αυτή την δυνατότητα επόμενο σημείο αφορά τα κολέγια. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι είναι περιτά και περίπλοκα. Κοιτάξτε, τα college υπάρχουν ήδη, λειτουργούν, είναι αποτελεσματικά και η μόνη χώρα που διαφωνεί είναι η Γερμανία. Εάν διαγράψουμε λοιπόν όλα αυτά τα κόλετζ από την πρόταση, χρειάζεται να κατανοήσετε πως η ΕΣΜΑ δεν αδειοδοτεί τα CCPs. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα college για να συνεργαστούν. Πρέπει να συμπεριλάβουμε τις κεντρικές τράπεζες στις συζητήσεις. Οι τροπολογίε του εισηγητή δεν ενισχύουν την ε, ΣΕΑΚΑ, δεν προβλέπουν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, αφήνουν το ζήτημα στα χέρια των εθνικών αρχών. ω εκ τούτου λοιπόν θέλουμε να υπάρχουν και να λειτουργούν αυτά τα κολέγια. Για τις τρίτες χώρες χρειάζεται να υπάρχει αμοιβαιότητα με αυτές. Ίσως να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς όρους, όχι η αμοιβαιότητα, όπως ισοτιμία. Εκεί που έχουμε σοβαρές ανησυχίες είναι τις προτάσεις που αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα των CCPs. Υπάρχουν μια σειρά τροπολογίες που ε, διαγράφουν ε, τα, το stress test ε, και λοιπά. Ας τα αφήσουμε αυτό στις διεθνείς μη δεσμευτικές ε, μη δεσμευτικούς κανονισμούς και ας διατηρήσουμε τους δεσμευτικούς για την Ευρώπη. Τέλος, η διαλειτουργικότητα. Είμαστε κατά της διαγραφής. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν ακριβείς ζητήματα, μόνο η Γερμανία και η Γαλλία είναι κατά αυτών. Δεν βλέπουμε συστημικά προβλήματα. Βλέπουμε κάποια ζητήματα τα οποία βελτιώνουν το μέρη, τα αγωνιστικότητα με αυτές τις χώρες ε, και αυτό το οποίο δεν επιθυμούν αυτές οι χώρες είναι ο ανταγωνισμός ε, και η ανταγωνιστικότητα. Η Κομισιόν λοιπόν ε, πιστεύει στην ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών αγορών και της ανταγωνιστικότητας στον τον κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Βέρνερ, εσύ. Ναι. Θα ήθελα να αρχίσω από το τέλος, από την Κομισιόν δηλαδή. Που βέβαια προασπίζεται και της πρόταση. Τα σχόλια όμως ήταν ένα μείγμα μεταξύ των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και αυτών που ακούστηκε εδώ. Για τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε μονάχα πώ θα συμφωνήσουμε μαζί με του στο τέλο. Όπως και ο κύριος και εγώ πιστεύω ότι για τα συντοξιδοτικά ταμεία, το είπε και συνάδελφος Φορτμαν Κόλ, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδική μορφή αναγνώρισης διμερών εκαθαρίσεων. Αυτό θα μπορούσε να ήταν κάποια εξαίρεση. Μετά, πεδίο εφαρμογή. Θα πρέπει να ρωτήσω τον υπεύθυνο υπάλληλο τη Κομισιόν. Μια που τα πράγματα είναι τώρα τόσο σαφή, γιατί δεν το πρότεινε η Κομισιόν έτσι. Και γιατί δεν το έλεγαν ούτε η ΕΠΑ υπόψη, ούτε οι, διασ... οι αποφάσεις της διάσκεψης κορυφής, ε, ούτε κανένα άλλος, θα συμπεριληφθούν όλα τα παράγωγα δηλαδή εδώ. Η Κομισιόν κάτι θα είδε που την έκανε να αλλάξει την άποψή τη. Εγώ βασίστηκα βέβαια στην πρόταση τη Κομισιόν. Αλλά αύριο έχουμε μια συνομιλία για το θέμα αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε. Για το backloading. Συμφωνώ με την άποψη που παρουσιάστηκε εδώ ότι υπάρχουν και νομικοί λόγοι, το έγραψα και στην εκδοσή μου, και ουσιαστικοί όμω επίση να μην έχουμε κανένα backloading, αλλά από τη στιγμή της θέση ισχύ ε, ε, του κανονισμού να υπάρχει η υποχρεώση αναφοράς. Κατόπιν. Ίσως εγώ δεν έχω τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν σε μια τηλεφωνική διάσκεψη. Αλλά έγινε μια ακρόαση, έχω το κείμενο εδώ που έχει σαν στόχο γίνεται μάλλον στην Αμερική αυτή τη στιγμή, όπου σε στόχο να εκτάσουν κατά πόσον μικρέ και μεσαίου ή μεγέθου τράπεζες μπορούν να έχουν μια γενική εξαίρεση από την υποχρέωση καθάρισης. και όχι όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, αλλά όσον αφορά το ποσό του ισολογισμού. Αυτό είναι διαφορετικό στις τράπεζες. Και αναφέρθηκε ένα τυχαίο αριθμό 10 δισεκατομμυρίων που θα πάρει κανένα οποιοδήποτε άλλο αριθμό ήθελε. Εγώ δεν προτείνω κάτι τέτοιο στη δική μου έκθεση και το υπέβαλα πραγματικά στις συζητήσεις γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η ακρόαση. Δεν έχω κάνει πρόταση, όλα είναι ανοιχτά προς το παρόν. Δεν θα πρέπει βέβαια να εργαστούμε εμείς εις βάρος των δικών μας μικρών τραπεζών. Το είδαμε με τη Βασιλεία 2. Επέμεινε η Κομισιόν να υιοθετήσουμε το γλυγορότερο δυνατόν την οδηγία δεν υπήρχε τίποτα για τις μικρομεσαίες τράπεζες και το αποτέλεσμα είναι ότι στη ΣΥΠΑ δεν επευλήθη κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα η δυνατότητα της αμοιβαιότητας να υπάρχει και να υπάρχει εξ αυτού και ε, προσαρμογή των εξαιρέσεων. Θα πρέπει να το ζητήσουμε. αλλά έχει δίκιο βέβαια ο κύριος Πίρσεν. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια αυστηρή διάταξη. Και παρεμβάσεις από εκείνους που συμμετέχουν στην αγορά είναι ότι δεν υπήρχε τίποτα, κανένα πολύ επικίνδυνο ο παράγωγο. Τώρα βέβαια εγώ θεωρώ τα δικά μου παράγωγα ότι δεν είναι επικίνδυνα του γείτονα. Ο γείτονα θεωρεί ότι τα δικά του δεν είναι επικίνδυνα του άλλου γείτονα. Λοιπόν, ο καθένα έχει λοιπόν μια επιθυμία πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ δεν προτείνω τίποτα. Μόνο στι αιτιολογικές σκέψει προσπάθησα να προβλέψω τι θα πρέπει να κάνει η ΕΑΚΑ και να υπάρχουν κάποιες σιγά σιγά διατάξεις. Τώρα για τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα συλλογικά σώματα, τα κολέγια, αποτελούν από δύο χώρες ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει η σύνθεση και το... η εντολή τους η σύνθεση είναι ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν πολλά μεγάλα παράγωγα δεν έχουν μια μεγάλη αγορά, δεν είναι κέντρο χρηματοπιστωτικό, ίσως δεν συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει όμως ότι οι μικρές χώρες ίσως ε, μπορούν να μπλοκάρουν ε, τους τρεις μεγάλους ε, τόπους χρηματοπιστωτικών κέντρων που έχουμε στην Ευρώπη. Εάν υπάρχει ευθύνη για την τελική δήλωση από τα συλλογικά αυτά στόματα κολέγια και όχι ΑΚΑ, βέβαια η ε, ΕΚΑ ίσως ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη στήριξη από τις εθνικές αυτές αρχές, αλλά το θέμα της έγκρισης και του ελέγχου στη χώρα ε, έγκρισης θα πρέπει να γίνεται από το εν λόγω κράτος μέλος. Αυτή η άδεια όμως θα είναι δυνατή μόνο μετά που θα υπάρχει γνωμοδότηση των συλλογικών οργάνων, των κολεγίων. Αυτό δεν μου φαίνεται όμως ότι είναι ισορροπημένο. Θα πρέπει να το ξαναμελετήσουμε κανονισμός για τις τρίτες χώρες και η διαλειτουργικότητα, η Κομισιόν προσανατολίστηκε και εγώ προσανατολίστηκα στο κείμενο της ε, ε Κομισιόν μόνο σε, ένα ορισμένο, μια ορισμένη μορφή των ε, παραγόγων αυτών. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα. Αλλά η γενική διεύρυνση της διαλειτουργικότητας μου φαίνεται πάρα πολύ προβληματική και ότι θα οδηγήσει σε μια αποδυνάμωση του συστήματος ή θα οδηγήσει σε συμπληρωματικούς κινδύνους του συστήματος και τελικά κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, ενδιαφέρομαι να έρθω σε επαφή και με την Κομισιόν και με τους αδέλφους εδώ στην Επιτροπή. Έχουμε μια καλή συνενετική και ισχυρή θέση τελικά και έναντι του Συμβουλίου. Γιατί το Συμβούλιο προσπαθεί από εδώ και επίσης τα ψηλά για να το πούμε έτσι, να διευρύνει τις αρμοδιότητές του. Για το σκιώδη συγητή των ε, Σοσιαλδημοκρατών, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή υποστήριξή σας όσον αφορά τις εξαιρέσεις, όσον αφορά την υποχρεώσια καθάρισης με τις 90 μέρες και τους 6 μήνες. Αυτή είναι η πρόταση βέβαια. Μπορούμε να τη διαπραγματευτούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να πούμε εάν μία μέρα ξεπερνάτε το επίπεδο εκαθάριση θα πρέπει αμέσως να υπάρχει συμπληρωματική ασφάλιση κλπ. κλπ. και Όλες αυτές τις υποχρεώσεις δηλαδή δεν μου φαίνεται ότι είναι σωστό. Κατά πόσα θα έχουμε μικρότερη διάρκεια, εντάξει αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όσον αφορά το κεφάλαιο είναι, είναι τυχαίο. Δηλαδή 5, δισεκατομμύρια, 10, δεν ξέρω αν θα αυτό αρκεί. Ίσως η Κομισιόν τη της εμπειρία να μπορεί να μας βοηθήσει. Κατόπιν, η κυρία Μπόλς αναφέρθηκε σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα που τα βλέπω κι εγώ έτσι όπως τα βλέπει εκείνη ιδίως οι δείκτες και η υποχρέωση αναφοράς που είναι διαφορετική από την υποχρέωση εκαθάρισης. Εάν έχουμε διαφάνεια κάτω των δυνατών και πρέπει να δηλωθούν όλες αυτές τις συμβάσεις, τότε οι εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τους κινδύνους ανεξάρτητα. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να, να περιοριστεί η υποχρέωση αναφοράς παρά μετά θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν πραγματικές υποχρεώσεις εκαθάρισης. Τι είναι κερδοσκοπικό. Δύσκολο αυτό. Κανένας δεν βρήκε λύση. Συζητιέται τώρα βάσει ενός ε, μη εγγράφου γαλλικού. Κάθε χώρα μέλος υποβάλλει τις δικές της ε, προτάσεις. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και ενδεχομένω και η Γερμανία έχουν διαφορετικά συμφέροντα από τη Μάλτα, η Κύπρος και η Λετωνία. Αυτονόητο αυτό. Γιατί αν δούμε το, τα δύο τρία της αγοράς ε, βρίσκονται στο Λονδίνο. Άρα θα πρέπει να εξαστούν τα επιχειρήματα που, βλέπω, που προέρχονται από εκεί. Κατά πόσο είναι βάσιμα. Είναι πιο σημαντικό παρά να εμπλακεί κάθε χώρα σε ένα σύστημα πληροφόρηση και αποφάσεις όταν δεν υπάρχει πραγματική σημασία για την αγορά. Πάντα σε αυτά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε λίγο πολύ. Ο Σάββας από τους πράσινους είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλικά πολλές εξαιρέσεις. Εγώ μία στιγμή ε, ε, δεν έχω προτείνει καμία εξαίρεση. Πολλές πολλές παρεμβάσεις που ακούστηκαν το είπα ρητά. Μόνο στις ετουλικές σκέψεις έχω ορίσει κάποιες υποχρεώσεις εξέτασης. Κυρία Σουίνπερν, όσον αφορά τα συνταξιδοτικά ταμεία, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είναι και ένα τμήμα του διακανονισμού που θα πρέπει να γίνεται από την ΕΚΑ οι κατηγορίες παραγωγών, οι διαφορετικές απαιτήσει, η δυνατότητα προστασία σε περίπτωση πτώχευσης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια κοινή λύση. Τελευταία παρατήρηση της Διευθυντικού Καταμία. Γιατί αυτό είναι κάπου που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Ολλανδούς που έχουν και διαφορετικά ταμεία από ότι άλλες χώρες ανά τον κόσμο Θεωρώ ότι οι παρατηρήσει είναι πάρα πολύ σωστές. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ μορφές collateral. Αυτό είναι κάτι που αφορά όχι μόνο τα κρατικά ταμεία, αλλά και τα, τα ταμεία επιχειρήσεων. Και υπάρχουν ορισμένε μεγάλε εταιρείε ε, στην Ευρώπη που έχουν τεράστια συνταξιδοτικά ταμεία και που θα τους ανέφερα το θέμα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προθεσμίες, ε, πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα. Προβλέπετο η 15η Μαρτίου. Σε δύο εβδομάδες, αλλά δεν αρχεί. 15 είναι Τρίτη, αν λέγαμε 17 ίσως θα είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν και κάποιες συνομιλίες πριν λύσει η προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τη ε, μετάφραση των εγγράφων αυτών, αλλά δεν έχουμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο βιάζεται, οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο. Τουλάχιστον αντί 15, ας παίρναμε την Τετάρτη το βράδυ, εάν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μου λέει η γραμματεία ότι ίσως έχουμε πρόβλημα αν προσπαθήσουμε να, προσπαθώντας να κάνουμε τις μεταφράσεις μια στιγμή. Το συζητήσουμε. Μετράμε τις μέρες. Γιατί πρέπει να έχετε και κάποιες μέρες στη διάθεσή σας για να υπάρχει μετάφραση, να έχουν μεταφραστεί τα κείμενα. Um, νομίζω ότι το επιβεβαιώνουμε. Σημειώνουμε λοιπόν ότι η συγητής ζήτησε να υπάρξει παράταση μέχρι Τετάρτη 17 ε, Μαρτίου η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, εφόσον τεχνικά είναι εφικτό. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. 16. Λοιπόν, βράδυ της 16ης. Καλώ. κάποιον θα σπρώξουμε κάπου για να το κρατήσουμε. Λοιπόν, βράδυ τη 16ης. Και 4 Απριλίου θα είναι η συζήτηση τροπολογιών με στόχο να γίνει σχετική ψηφοφορία 20 Απριλίου. Τώρα στα διάφορα δεν έχω τίποτα να προσθέσω και αυτό λεχθέντον λίγη τη συνεδρίαση.